and has made a real impact since its launch in. two thousand and seven i would like to thank you for giving me this opportunity to present the communication. θα ήθελα να δραχθώ της ευκαιρίας ώστε αυτή την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να την παρουσιάσω σε σχέση με την επικέντρωση και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας στην καινοτομία και την έρευνα. Αυτή η ανακοίνωση προτείνει μια νέα στρατηγική για τη διεθνή συνεργασία. Οι επιστήμονες πάντα περνούσαν τα σύνορα για να δώσουν συνέχεια στις ανακαλύψεις τους και συνεργαζόντουσαν με τους ομολόγους τους σε άλλες χώρες για να πετύχουν νέες ευκαιρίες. Ενώ αυτό ίσχυε για πολλούς αιώνες, ακόμα περισσότερο ισχύει σήμερα την εποχή της παγκόσμιας επικοινωνίας και αλληλεξάρτησης. Αυτό που βιώσαμε ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία είναι η δημιουργία ενός παγκόσμιου τοπίου όπου οι επιστημονικές δημοσιεύσεις όλο και περισσότερο συντάσσονται από ερευνητές διαφορετικών χωρών. Βλέπουμε επίσης αυτή την παγκοσμιοποίηση και στον ιδιωτικό τομέα εξίσου. Είναι Ευρω... ε, παγκόσμιος προπομπός πρωτοπόρος η Ευρώπη, ενώ η Ευρώπη είναι μόνο το 7% του παγκόσμιου πληθυσμού. Είναι υπεύθυνη όμως για 24% των παγκόσμιων δαπανών για την έρευνα. 32% των υψηλού επίπεδου δημοσιευμάτων και μεγαλύτερο ποσοστό ακόμα όσον αφορά τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Με το παγκοσμιοποιημένο τοπίο για την έρευνα βλέπουμε ότι πολλές νέες χώρες, οι χώρες BRIC, Βραζιλία, Ρωσία, Κίνα, Ινδία, επενδύουν σε σημαντικότατα, με σημαντικότατα ποσά για προγράμματα και σχέδια έρευνας. Αυτές οι τάσεις είναι προκλήσεις και ευκαιρίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση ταυτόχρονα. Η γνώση γεννάται εκτός Ευρώπης και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι δικοί μας ερευνητές και οι δικές μας επιχειρήσεις θα έχουν πρόσβαση σε αυτή τη γνώση. Παγκοσμιοποίηση και κινητοποίηση, κινητικότητα οδήγησαν σε ένα νέο τοπίο για τον ανταγωνισμό μεταξύ των ταλαντούχων. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα κλιματολογικές προκλήσεις, ε, η διάδοση μολυσματικών ασθενειών, ε, η διασφάλιση των ενεργειακών μας αναγκών με καθαρή ενέργεια απαιτεί να συνεργάζονται οι επιστήμονες με τον καλύτερο τρόπο για να εξεύρουν λύσεις σε αυτά τα παγκόσμια προβλήματα και προκλήσεις. Σε συνεργασία με τους εταίρους μας μπορούμε να βρούμε τις απαντήσεις και να δημιουργήσουμε μίζονες ευκαιρίες ε, για, ευκαιρίες για να μπορέσει να υπάρξει αυτή η ανάπτυξη. Είναι λοιπόν σημαντικότατο. Η διεθνής αυτή συνεργασία πρέπει να εξακολουθήσει να είναι θεμελιώδης λίθος της πολιτικής μας και θα πρέπει να είναι και ένα από τα κυριότερα στοιχεία του ορίζοντα 2020. Αυτή η νέα στρατηγική θεμελιώνει στα επιτεύγματα του 7ου προγράμματος πλαισίου. Υπάρχουν πολλά καλά παραδείγματα, ας αναφέρω κάποια από αυτά. Το 7ο πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης οδήγησε ε, στην ανάπτυξη εταιρική σχέσης όπου 14 κράτη-μέλη και η Νορβηγία και η Ελβετία συνεργάστηκαν με υποσαχάριες ε, στη μεσημβρινή Αφρική χώρες για να καταπολεμηθεί το AIDS, η ελονοσία, η... Ε, θυματίωση. Συμμετείχαν όλες αυτές οι χώρες ε, στην Μαρίς Κλοντόφσκα Κουρί δράση στις δράσεις αυτές έτσι οι αν, ανώτατου επίπεδου επιστήμονες οπουδήποτε και αν βρίσκονται μπορούν να διεξάγουν αυτή την, διεξάγουν την έρευνα στην Ευρώπη. Με αυτή την αλληλεξάρτηση και διασύνδεση των θεσμικών οργάνων που επικεντρώνονται και στην Ευρώπη χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο, 7ο Πλαίσιο για την Έρευνα και την Ανάπτυξη. Το σχέδιο ITER αποκινούμε την Κίνα, η Ιαπωνία, ΗΠΑ, Ρωσία, Ινδία και Νότια Κορέα Προσπαθούμε να καταδείξουμε την βιωσιμότητα της ε, ε, ε, πυρηνικής σύνδεξης και αυτό είναι μια ναυαρχίδα όσον αφορά τις διεθνείς μας συμφωνίες ε, και προγράμματα και σχέδια. Κάνοντας τόσο μεγάλα βήματα στη διεθνή συνεργασία, καθίσταται σαφές ότι πολλά ακόμα πρέπει να γίνουν. Προς αυτόν τον στόχο η νέα στρατηγική μας έχει τρεις κύριους άξονες ως στόχους. Πρώτον, να εντείνουμε και να ενισχύσουμε την βελτιστή πολιτική για την αριστεία από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να αποκομίσει τα μέγιστα ωφέλη η Ευρώπη, πρέπει να έχουμε πρόσβαση στη γνώση, στου κατάλληλου τους ανθρώπους και στις αγορές παγκόσμια. Δεν είναι όμως μονόδρομος αυτή η πορεία. Για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε αποτελεσματικά πρέπει να διασφαλίσουμε ότι επίσης θα παραμείνουμε ελκυστικός, θελκτικός εταίρος παγκόσμια. Δεύτερον, αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων. Πρέπει παγκόσμια να συνεργαστούμε για να αντιμετωπιστούν οι κυριότερες κοινωνικές προκλήσεις στις οποίες προαναφέρθηκα. Τρίτον, να υποστηρίξουμε τις ε, εξωτερικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλές από τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που προσυπογράψαμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτές πάλι από την έρευνα και την ε, ανάπτυξη χαρακτηρίζονται. Δεσμεύσεις μας στην περιοχή της Λεκάνης της Μεσογείου αλλά και άλλες διεθνείς υποχρεώσεις και δεσμεύσεις. Η επίτευξη των στόχων της χιλιετίας, η δέσμευσή μας να υποστηρίξουμε αναπτυσσόμενες χώρες να αναπτύξουν τις κοινωνίες και τις οικονομίες τους. Ορίζοντας 2020 θα ξεκινήσει ως πρωτοβουλία το 2014. Θα είναι το κυριότερο μέσο ως εργαλείο για να επιτύχουμε την διεθνή αυτή μας συνεργασία. Διτή προσέγγιση θα υιοθετηθεί. Πρώτον, ορίζοντας 2020 θα είναι ανοιχτός για την συμμετοχή από όλες τις χώρες, επιτρέποντας σε κονσόρτσια της Ευρώπης να συνεργάζονται με ομόλογους και εταίρους παγκόσμια σε θέματα που θα επιλέγουν. Δεύτερον, θα έχουμε στοχοθετημένες δράσεις, ε, όπου εμείς ως υπεύθυνοι για τα πολιτικά θέματα θα αποφασίζουμε εκ προηγουμένου ποια θα είναι η περιοχή, το πεδίο έρευνας και ποιοι οι ομόλογοι μας, οι εταίροι μας. Θα επιλέγονται με βάση κοινά συμφέροντα και κοινό όφελος όλα αυτά. Θα αναπτύσσονται από τον σε εξέλιξη διάλογο με τους παγκοσμίου, παγκόσμιους εταίρους μας. Ορίζοντας 2020 θα αποτελέσει σημαντική βελτίωση, διασφαλίζοντας μια στρατηγική, πιο στρατηγική προσέγγιση για αυτούς τους στόχους, με επιλογή που θα βασίζεται σε σαφέστατα κριτήρια μέσα σε ένα συνεκτικό πλαίσιο για το σύνολο του προγράμματος. Επίσης θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας να αναπτυχθούν δράσεις σε επαρκή κλίμακα και εμβέλεια ώστε να υπάρξει η αναγκαία επίπτωση ως αποτέλεσμα όπως επιθυμούμε. Όλα αυτά θα εξηγούνται σε μια σειρά οδικών χαρτών που θα επεξηγούν για ποιες χώρες, περιφέρειες, ομολόγους εταίρους μας και για ποια θέματα θα υπάρχει αυτή η συνεργασία στην έρευνα, ώστε οι ερευνητές μας να μπορούν σε ένα πλαίσιο αμοιβαία εμπιστοσύνη να συνεργάζονται με τους ομολόγους τους παγκόσμια. Γι' αυτό χρειάζεται ένα ισοδίκαιο πλαίσιο ισότιμης συμμετοχής. Η στρατηγική λοιπόν αυτή προάγει την προώθηση κοινών αρχών και θεμελίων στα διεθνή αυτά ζητήματα για την έρευνα, κεραιότητα, φύλλο, αμοιβαιότητα και ανοιχτή πρόσβαση και προσπελασιμότητα η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων θα είναι μεγάλη σημασία για τον ορίζοντα 2020 και για την μεγάλη σημασία για τις δραστηριότητες καινοτομία. Η στρατηγική αυτή δεσμεύει και φέρνει πιο κοντά για τις πολιτικές αυτές και την χρηματοδότηση των προγραμμάτων αυτών τα κράτη-μέλη μας με άλλους εκμεταλλευόμενοι ιδιαίτερα το Φόρουμ για τη Διεθνή Επιστήμη και την Τεχνολογική Συνεργασία. Αυτό το θεσμικό όργανο συνενώνει τα κράτη-μέλη, τις χώρες που συνδέονται με το πρόγραμμα πλαίσιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόσφατα, τα τελευταία χρόνια, αυτό το φόρουμ, αυτό το βήμα ανέπτυξε συγκεκριμένα θεματολόγια ως ημερήσιες διατάξεις με χώρες κυρία σημασίας όπως την Ινδία, την Βραζιλία, τη ΣΥΠΑ, την Κίνα. Πρέπει να συνεχίσουμε να δίνουμε αυτή την προώθηση και να προάγουμε όλα αυτά τα θέματα. Ξεκίνησαν προσπάθειες για την εκμετάλλευση καλύτερων συνεργειών και σχέσεων μεταξύ εθνικών και διεθνών προγραμμάτων, δίνοντας τη δυνατότητα να υπάρχουν περισσότερο διεθνοποιημένα τέτοια προγράμματα. Η καθέλκυση, η εκκίνηση αυτής της στρατηγικής είναι μόνο το πρώτο βήμα. Για να μπορέσει να λειτουργήσει θα απαιτηθεί η ευδιάκριτη συνεργασία σε πλήρη βαθμό στον ε, ορίζοντα 2020. Για να διασφαλίσουμε ότι θα παραμείνουμε σε αυτή την πορεία και τροχιά θα υποβάλει αναδιετή διαστήματα έκθεση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μετράτε η πρόοδος και να αξιολογείτε το κεκτημένο και τα επιτεύγματα. Είναι τεράστια σημασία σε όλα αυτά για να μπορέσουμε να δρέψουμε τους καρπούς από αυτή τη διεθνή συνεργασία στην έρευνα και να έχουμε αυτή την πρωτο... αυτό τον ρόλο που είναι πραγματική δική μας πρωτοβουλία. Θα πρέπει να έχει τεράστια σημασία για την επίτευξη των στόχων μας. Ευχαριστώ. Grazie al commissario per il suo intervento. Iniziamo subito il dibattito dando la parola alla collega Carvaio. Prego. Thank you, President Sartori. I would like to congratulate and welcome the Commissioner again to our committee. Ήθελα να συγχαρώ την Επιτροπή για το ότι έκανε μια πάρα πολύ καλή ανακοίνωση, μια ανακοίνωση που ήταν απαραίτητη, διότι κατά το παρελθόν ε, δεν είχαμε την <clears throat> στρατηγική προσέγγιση στη διεθνή συνεργασία. Επίσης, ε, δεν ε, μπορέσαμε να επεκταθούμε όσον αφορά την ε, διεθνή συνεργασία. Μερικές φορές υπάρχει ένα ξεχωριστό πρόγραμμα για τη διεθνή συνεργασία με ορισμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Άλλες ε, φορές πάλι οι απόψεις αυτές διεισδύουν σε διάφορα υποπρογράμματα και διάφορες προτεραιότητες. Πάντως, ποτέ δεν υπήρξε ή δεν αναφέρθηκε ότι η στρατηγική είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστεί η διεθνή συνεργασία. Είναι λοιπόν ιδιαίτερα ευχάριστο το γεγονός ότι υπάρχει τώρα αυτή η στρατηγική που περιλαμβάνει τη διεθνή συνεργασία για την έρευνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω την ε, υποστήριξή μου σε δύο θέματα. Στο θέμα της συμμετοχής διαφόρων κρατών, φαντάζομαι ε, η Πίτροπος δεν το είπε, αλλά το υποθέτω ότι όσον αφορά τις μορφές ε, καταβολής αυτό θα ε, συμπεριληφθεί ε, στον, στη συμφωνία περί συμμετοχής. Εκεί θα οριστούν οι λεπτομέρειες για το πώς θα συμμετέχουν οι διάφορες χώρες στους μηχανισμούς χρηματοδότησης. Αυτό είναι η πρώτη μου ερώτηση. Και παράλληλα υπάρχει και μια άλλη προσέγγιση που είναι τα μέτρα στόχος. Νομίζω ότι είναι ε, σημαντικό να υπάρχουν ε, μέτρα στόχος ε, όπως η φτώχεια που έχει σχέση με τις ασθένειες στην Αφρική ή τα βιοκάψιμα στη Βραζιλία. Αυτή είναι, αυτές είναι στοχευμένες ενέργειες για συγκεκριμένες χώρες. Στην ανακοίνωσή σας αναφέρεται ότι θα υπάρξουν πολιτείς χάρτες πορείες σχετικά με τη συνεργασία. Και η τελευταία ερώτηση που υποβάλλω εγώ είναι η εξής. Υπάρχει ένα πολύ σφιχτό χρονοδιάγραμμα, έτσι ώστε οι χάρτες αυτή πορείας να είναι αποτελεσματικοί ε, στον ορίζοντα 2020. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό ε, όταν θα ξεκινήσει το πρόγραμμα ορίζον ε, το 2014, τότε να γνωρίζουμε πολύ καλά τους ε, χάρτες πορείας, τους στόχους ε, που θα υπάρχουν σχετικά με τη συνεργασία. Και ρωτώ, ε, εσείς πώς βλέπετε να, είναι, να υπάρχει συμβατότητα ανάμεσα στα δικά σας τα προγράμματα και στο πρόγραμμα Horizon 2020. Τέτοιου είδους χάρτες πορείας θα υπάρξουν στο τέλος του 2013 έτσι ώστε το 2014 να μπορούμε να ξεκινήσουμε με την, ε, τη συνεργασία, τη στοχευμένη συνεργασία με τους στρατηγικούς μας εταίρους. Ευχαριστώ πολύ. Η συνάδελφος Ριέρα Μαντουρέλ, παρακαλώ. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, καλώ ήρθατε. Επίση και εξ ονόματο τη ομάδα μου σε αυτήν την Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Και όπω πάντα, σα ευχαριστώ και ε, σας ευχαριστούμε για αυτή την παρουσία σας ενώπιόν μας. Και εγώ περισσότερο από ερώτηση θα ήθελα ένα σύντομο σχόλιο να κάνω. Και επίσης συσχετίζεται αυτό κυρίως με τη σχέση της ανακοίνωσης που μας παρουσιάσατε με το νέο πρόγραμμα πλαίσιο Οριζόντα 2020 όπου όπως πολύ καλά γνωρίζετε η δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή εργάζεται εργοδός με έντονους ρυθμούς. Η ομάδα μου είναι πεισμένη ευθύ εξ αρχής για την ανάγκη να προχωρήσουμε στην οικοδόμηση αυτής της Ευρώπης και για αυτόν τον ορίζοντα και την έρευνα και την ανάπτυξη. Και για να πετύχουμε αυτό πρέπει να αναπτύξουμε τη διεθνή διάσταση της έρευνας και ανάπτυξης και συνεργασίας. Είναι προφανές επιπλέον ότι η Ευρώπη σε αυτή τη χρονική συγκυρία μπορεί να απαντήσει πιο αποτελεσματικά στην πλειοψηφία των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας μέσα από το πλαίσιο της στρατηγικής 2020 για την ε, ενεργειακή κάλυψη των αναγκών μας και άλλων ε, τέτοιων στόχων που είναι παγκοσμιοποιημένοι με μεγαλύτερη ολοκλήρωση και συντονισμό των δράσεων στην έρευνα και την καινοτομία πέρα από τα σύνορά μας και να συνεχίσουμε να προαγάγουμε την τεχνολογική συνεργασία και επιστημονική συνεργασία με τρίτες χώρες. Για όλους αυτούς τους λόγους πιστεύουμε και θεωρούμε ότι το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 πρέπει να αντανακλά με σαφήνεια, με σαφή τρόπο αυτή την ανάγκη. Εσείς σήμερα με σαφή τρόπο το εξηγήσατε. Πρέπει αποτελεσματικά να έχουμε αυτό το πρόγραμμα για τη συνεργασία με τρίτες χώρες στην έρευνα και ανάπτυξη. Όμως ουσιαστικά στην πρόταση που ήρθε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Ευρωκοινοβούλιο την πρόταση για το πρόγραμμα αυτό, η ομάδα μας θεώρησε ότι αυτό το θέμα ούτε επαρκώς δεν είχε αποσαφινιστεί, ούτε επαρκώς είχε αναπτυχθεί. Και γι' αυτό πρέπει να πω ότι μας παραξένεψε αυτό στη συνέχεια, διότι συμμεριζόμαστε όλα τα όσα είπατε σήμερα ενώπιόν μας. Τα συμμεριζόμαστε απόλυτα. Και γι' αυτό <laughs> σε σχέση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η ομάδα μας θεώρησε σημαντικό να καταθέσει μια τροπολογία λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα οποία μάθαμε από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, όπως πολύ καλά είπατε, κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης και εκτέλεσης αυτού του 7ου προγράμματος πλαισίου. Καταθέσαμε λοιπόν μια τροπολογία όπου υπογραμμίζαμε την ανάγκη να βελτιωθούν και να γίνουν πιο αποτελεσματικά τα αναγκαία μέτρα και εργαλεία ώστε να υπάρχει μια πιο αποτελεσματική συνεργασία σε παγκόσμια κλίμακα που είναι τόσο αναγκαία. Και εγώ θα ήθελα επίσης να πω, είναι με βεβαία ότι γνωρίζετε την τροπολογία μας, θα ήθελα να μου πείτε κάπως ποια είναι η άποψή σας για αυτή την τροπολογία μας. Και τι σκέφτεστε για όλα αυτά τα οποία τότε στο παρελθόν κάπως μας είχαν παραξενέψει. Μια και αυτό είναι το περιεχόμενο της τροπολογίας μας, η διεθνή συνεργασία πρέπει να είναι διπλή κατεύθυνσης. Όπως πολύ καλά εξηγήσατε, αφενός πρέπει να προχωρήσουμε στην επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία με τα πιο προηγμένα κέντρα παγκόσμια. Πράγμα που θα μας βελτιώσει, δώσει την δυνατότητα να βελτιώσουμε την αριστεία μας και να ανταγωνιστούμε στο μεγαλύτερο, ανώτερο, υψηλότερο επίπεδο. Αλλά επίσης σκεφτόμαστε ότι πρέπει να προχωρήσουμε στην τεχνολογική και επιστημονική συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες εκμεταλλευόμενοι όλο το δυναμικό της καινοτομίας και της επιστήμης για να παγιωθούν ευάλωτες κοινωνίες και να συνεισφέρουμε έτσι υπέρ της ειρήνης και της παγκόσμιας σταθερότητας στη σταθεροποίηση αυτή. Γι' αυτό, Επίτροπε, η πρόταση η οποία θα διατυπωθεί από το Κοινοβούλιο σε σχέση με αυτό το πρόγραμμα, την πρόταση Ορίζοντα 2020, θα πρέπει να ενισχυθεί η διεθνή συνεργασία διότι συμφωνούμε. Είναι ένα καλό μέσο και εργαλείο για να ενισχύσουμε το σύστημά μας έρευνας και ανάπτυξης. Και πιο πριν αναφέρατε την βελτίωση του πλαισίου αριστείας, αλλά είναι επίσης ένα θετικό καλό μέτρο για να έρθουμε σε επαφή με τους καλύτερους ερευνητές και ερευνητικά κέντρα τρίτων χωρών και να προσελκύσουμε, να θέλξουμε τους πιο ταλαντούχους, ώστε να υπάρξουν και επενδύσεις που θα διασφαλιστούν, να διευκολυνθεί η πρόσβαση στις νέες αγορές, να βελτιστοποιηθούν οι χρήσει των υποδομών, στην έρευνα κτλ. Είναι ένα λοιπόν πολύ καλό μέσο αυτό. Εξαιρετικό μέσο θα έλεγα, εξαίσιο μέτρο και εργαλείο για να βελτιώσουμε το σύστημα στην έρευνα και ανάπτυξη. Είναι ένα καλό μέσο, όπω είπα, όπω αναφέρθηκε, για να αντιμετωπιστούν οι παγκόσμιες προκλήσεις, που παγκόσμια, παγκοσμιοποιημένα πρέπει να αντιμετωπιστούν και να εκπονήσουμε πολιτικέ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω την πολιτική ασφάλεια, την ενεργειακή μα πολιτική, την πολιτική μα για την συνεργασία στην ανάπτυξη. Γι' αυτό θα ήθελα να κάνω λοιπόν αυτό το σχόλιο, Επίτροπε, σε σχέση με το πώ προσεγγίσαμε αυτό το θέμα μέσα στο πρόγραμμα πλαίσιο που σίγουρα θεωρήσαμε σε σχέση με το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο ότι είχε λιγότερο αναπτυχθεί. Τώρα μας καθησυχάσατε με την παρέμβασή σας και παρουσία σας και με αυτά που είπατε. Και προσθέτω τη φωνή μου στα σχόλια της κυρίας Καρβάλιο για το έφθετο αυτής της ευκαιρίας, ώστε να μην υπάρχουν αμφιβολίες. Να αρθούν όποιες αμφιβολίες υπάρχουν για αυτό το θέμα το οποίο είναι τόσο σημαντικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, συνάδελφος Τικάου, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επίτροπο για την έλευσή της εδώ, ενώπιον μας, σήμερα. Και θα ήθελα να τονίσω την σημασία της έρευνας και της για την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, η σημασία της τεχνολογίας και της καινοτομίας είναι εξαιρετικά σημαντική. Για να υπάρξει ανταγωνιστική βιομηχανία, χρειαζόμαστε πόρους, φυσικούς πόρους, αλλά και αποδοτική χρήση των πόρων. Για το λόγο αυτό θεωρώ ότι είναι σημαντική η διεθνή συνεργασία σε τρόπο ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει να αναπτύξει έρευνα και καινοτομία με στόχο την αποδοτική χρήση των φυσικών πόρων και κυρίως για τον εξυγχρονισμό της ευρωπαϊκής βιομηχανίας έτσι ώστε να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να παραμείνει ανταγωνιστική στο διεθνές επίπεδο. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα στα διεθνή πλαίσια είναι σημαντική και νομίζω ότι είναι επίσης σημαντικό μέσα στα πλαίσια αυτά, μέσα σημαντική μάλλον στα πλαίσια αυτά, η διαστημική έρευνα. Εκεί είναι ουσιώδης η διεθνή συνεργασία. Το πρόγραμμα Γαλιλαίος είναι ένα σημαντικό έργο και η παρατήρηση της γης από το διάστημα καθώς και άλλοι τομείς της έρευνας που έχουν σχέση με το διάστημα μπορούν να γίνουν και σε διεθνές επίπεδο. Το ίδιο για την πυρηνική ενέργεια, που είναι τομέας ο οποίος απαιτεί ε, αυξημένη, ενισχυμένη διεθνή συνεργασία. Εν τέλει, δε, κυρία Επίτροπε, είναι πολύ σημαντικό να γίνουν περισσότερα, να επενδυθούν περισσότερα ώστε οι δημοσιεύσεις που είναι γνωστές στον επιστημονικό κόσμο να μπορέσουν να διαδοθούν περισσότερο στην ευρωπαϊκή επικράτεια. Χρειαζόμαστε καλύτερες δημοσιεύσεις στον τομέα της έρευνας και αυτό το βήμα νομίζω θα προσφέρει κίνητρα σε νεαρούς ερευνητές να συνεχίσουν τις έρευνές τους στους τομείς αυτούς. Εύχομαι στη στρατηγική που θα προωθήσετε να δώσετε περισσότερο χώρο στην διαστημική έρευνα, στην πυρηνική ενέργεια και στη βιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χωρίς επενδύσεις δεν θα έχουμε ποτέ ανταγωνιστική βιομηχανία. Ευχαριστώ. Κρόλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε και την Επίτροπο σήμερα που ήρθε εδώ κοντά μα. Ε, κύριε Επίτροπε, θα γνωρίζετε πολύ καλά ότι εμεί σα στηρίζουμε ανεπιφύλακτα ε, όσον αφορά στο ρόλο και τη σημασία τη έρευνα και τη ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και γενικότερα στον κόσμο. Επιθυμούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρίσκεται στην αιχμή του δόρατο στην ε, έρευνα. Ε, τρία πράγματα με απασχολούν. Πρώτον, τα κονδύλια. Πόσα χρήματα μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι στο μέλλον θα προβλέπονται στον προεπλογισμό για μας. Δεύτερον, πολύ σύντομα, δείξατε το θέμα της ε, πνευματικής ε, ιδιοκτησίας και των ιδεών που απορρέουν από την έρευνα και κυρίως ε, από την έρευνα μέσα από τη συνεργασία. Κατά το παρελθόν κάναμε την εμπειρία ότι πολλές μορφές συνεργασίας στο, για το iPad και το iPhone. Ε, αυτά ξεκίνησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως τελικά τα εκμεταλλεύτηκαν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Ε, ξέρω ότι αυτό δεν είναι δικό σας τομέας, όμως οι συνάδελφοί σας, οι επίτροποι, αυτοί τι ακριβώς ρόλο ε, διαδραματίζουν σχετικά με, την, με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Όσον αφορά τις γραφειοκρατικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι υπάλληλοι τους που θέλουν να ασχοληθούν με την έρευνα, αλλά δεν έχουν ούτε το χρόνο ούτε τη δυνατότητα ε, που έχουν αυτοί που εργάζονται σε μεγάλες πολυεθνικές. Ίσως λοιπόν θα πρέπει κανείς να το σκεφτεί αυτό, αυτές τις ομάδες ε, να μπορούν και αυτοί οι άνθρωποι να εργαστούν όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε υπερεθνικό επίπεδο. Και τέλος όσον αφορά την πρόσβαση ε, στους ανθρώπους. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Να μπορείτε να φέρετε πιο κοντά ανθρώπους με διαφορετικές ειδικότητε, να συντονίζετε η δουλειά τους, γιατί όταν μιλάμε για ανθρώπους, ε, δυστυχώς ξεχνάμε ότι πολλές φορές μιλάμε για επαΐοντες που γνωρίζουν άλλους ειδικού, αλλά δεν γίνεται σωστή εκμετάλλευση των γνωριμιών. Ίσως θα μπορούσαμε αυτούς τους ανθρώπους να τους φέρουμε πιο κοντά σε ομάδες και με τον τρόπο αυτό θα μπορούσαν και αυτοί να μοχλεύσουν χρήματα από την οικονομία και έτσι να δώσουν μεγαλύτερη σημασία στην έρευνα και την ανάπτυξη. Και τέλος, αναφερθήκατε στα, ε, στους πολιτείς χάρτες πορείας. Πιστεύετε ότι μέσα από αυτούς τους χάρτες μετά από δύο χρόνια θα μπορεί κανείς να επιτύχει τα αποτελέσματα που είναι απαραίτητα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο συνάδελφος Τόμψεν έχει το λόγο. Ή κυρία Τόμψεν, με συγχωρείτε. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε που ήρθατε σήμερα εδώ και θα ήθελα επίση ε, να σας ε, συγχαρώ όσον αφορά αυτή η στρατηγική προσέγγιση για τη διεθνή συνεργασία. Δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο το γεγονός ότι κατατείται τώρα αυτή η πρόταση, γιατί τώρα ε, υπάρχει η παγκοσμιοποίηση και όλες οι χώρες αρχίζουν πια να συνεργάζονται. στη συνάντηση στο συνέδριο που έγινε στο Δουβλίνο πληροφορήθηκα ότι υπάρχει μία μορφή συνεργασία Βραζιλία, Νότιο Αφρική, Ινδία. Ε, σε αυτές τις χώρες οι επιστήμονες μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα και η ιδέα είναι ε, να έχουν ε, την επιστήμη χωρίς σύνορα. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί, οι επιστήμονες, θα μπορούν να μετακινούνται ελεύθερα τόσο οι επιστήμονες όσο και οι φοιτητές. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω σε εμά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη συνεργασία που έχουμε με τρίτες χώρες, είπατε ότι το δεύτερο ε, σημαντικότερο είναι να αντιμετωπίσει κανείς αυτές τις ε, παγκόσμιες ε, προκλήσεις έτσι ώστε να προσελκύσει τα καλύτερα ταλέντα. Μπορώ λοιπόν να φανταστώ ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα υπάρξει κάποια σύγκρουση. Βλέπω ότι ορισμένες χώρες είναι περισσότερο προστατευτικές από άλλες και εμείς τελικά χρηματοδοτούμε τους καλύτερους Αμερικανούς για να έρθουν εδώ να αποκτήσουν γνώση για την Ευρώπη. Θα ήθελα λοιπόν να ενημερωθώ λιγάκι και για τη χρηματοδότηση. Ποιο καλείται να, να χρηματοδοτήσει τη συνεργασία με τις ε, τρίτες χώρες και τι συμβαίνει με την ανταλλαγή φοιτητών από τρίτες χώρες. Ε, αυτό πώς μπορεί ακριβώς ε, να οργανωθεί. Αυτά είναι τα ερωτήματα που είχα να σας απευθύνω. Κοσέ έχει το λόγο. Επόμενος, ο κύριος Κοσέ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και ευχαριστώ βεβαίως και την κυρία Επίτροπο για τις δηλώσεις της. Με την ευκαιρία δε συγχαίρω και τον συμπατριώτη μας Σέρς για το βραβείο Νόμπελ που έλαβε σήμερα. Διεθνή συνεργασία και το πρόγραμμα και οι προσανατολισμοί του ορίζοντος 2020 εκπλήσουν διότι όπως είπε και η συνάδελφός μου εδώ αριστερά το μεγαλύτερο μέρος των ενισχύσεων δίνονται για έργα υψηλής τεχνολογίας, high-tech δηλαδή που χρησιμοποιούν πρώτες ύλες που έρχονται από όλο τον κόσμο και που εξ αντιθέτου όταν επιθυμεί κανείς να αναπτύξει συνεργασία με ορισμένες άλλες χώρες ιδίως του νότιου ημισφαιρίου δεν είναι ίσως η πρώτη τους προτεραιότητα. Αγαπητοί συνάδελφοι, μιλήσατε για την πυρηνική ενέργεια και την αεροναυτική. Ειδικώ για την πυρηνική ενέργεια δεν νομίζω ότι είναι βιομηχανία του μέλλοντος. Βεβαίως αυτά είναι αποφάσεις χαρακτήρως πολιτικού, εάν δηλαδή θα ενισχυθεί περισσότερο μία συνεργασία και όχι μία άλλη. Εγώ πάντως θεωρώ ότι σε συνεργασία με όλες τις χώρες του κόσμου και εδώ είναι το ερώτημα που θέτω στην κυρία Επίτροπο, μήπως πρέπει να αναζητήσουμε πολύ στοχευμένες και επιστημονικές συνεργασίες χαμηλής τεχνολογίας, ας πούμε low-tech, για να δημιουργηθούν προϊόντα τα οποία είναι, είναι χρήσιμα για κόσμο που δεν έχει, καθημερινά δηλαδή, για κόσμο που δεν έχει στη διάθεσή του ηλεκτρικό ρεύμα. Διότι μιλούμε για εκατοντάδε εκατομμύρια ανθρώπων που δεν μπορεί να επωφεληθεί από, μια, από, από ένα ηλεκτρικό πλυντήριο διότι δεν έχει ηλεκτρικό ρεύμα. Μπορεί όμως να πλύνει τα ρούχα του διαφορετικά. Ή για την γεωργία, την διαρκή βιώσιμη καλλιέργεια που είναι χαμηλής τεχνολογίας αλλά πολύ επιστημονική. Βλέπει Νότια Αμερική και Αυστραλία, που δεν τη βλέπω όμω στα προγράμματα του ορίζοντο 2020. Τελειώνοντας, κυρία Επίτροπε, δεν νομίζετε ότι για να ανταποκριθούμε στι ανάγκε ορισμένων τμήματων πληθυσμού του Νότιου ημισφαιρίου θα χρειαστεί μια πολύ σοβαρή επιστημονική συνεργασία, αλλά ξαναλέω low-tech. Ευχαριστώ. Ας Ευχαριστώ πρόεδρε. Θέλω να χαιρετήσω θερμά την κυρία Επίτροπο και να υπογραμμίσω και να πω ότι αυτή η στρατηγική εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν αναγκαία και χαιρετίζουμε όλοι μας αυτή τη στρατηγική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια ιδιότητα όσον αφορά την έρευνα. Είναι μια νησίδα έρευνα ας το πω έτσι. Και γι' αυτό είναι δύσκολο να υλοποιηθεί μια τέτοιου είδους συνεργασία και να επιτευχθεί ένας τέτοιος συντονισμός. Και όσο αφορά την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, πάλι δεν βρισκόμαστε σε ένα ενιαίο πλαίσιο όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν άλλα πεδία και θέματα όπου έχουμε προχωρήσει πιο πολύ. Ένα ενιαίο σύστημα ε, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας θα μας δώσει τη δυνατότητα αυτό, τις διάσπαρτες ε, δυνατότητες που έχουμε, το διάχυτο δυναμικό μας να το συνενώσουμε και να το καταστήσουμε πιο αποτελεσματικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι λοιπόν ένα ιδιαίτερο μόρφωμα, ένα ιδιαίτερο δημιούργημα σε σχέση με τα κράτη-μέλη και την Ένωσή τους. Υπάρχουν μεταξύ των διαφορετικών κρατών μελών διαφορετικά πανεπιστήμια. Πρέπει να πετύχουμε μια συνέργεια αποτελεσματική μεταξύ των κρατών μελών, των ερευνητικών ιδρυμάτων, των πανεπιστήμιων πανεπιστημίων για να μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε παγκόσμια όσον αφορά τα ευρωπαϊκά, το Ευρωπαϊκό Τεχνολογικό Ίδρυμα και το, το Ίδρυμα για την Καινοτομία θα ήταν ένα σωστό βήμα προς την αυτή, σωστή κατεύθυνση. Άλλα βήματα πρέπει να ακολουθήσουν μετά οπωσδήποτε. Θέλω να ερωτήσω την κυρία Επίτροπο. Έχει υπόψη της ε, τέτοιου είδους ιδρύματα και θεσμικά όργανα να τα δημιουργήσει και να τα προαγάγει. Θα χρειαζόμαστε τέτοια ενιαία ιδρύματα και θεσμικά όργανα. Κατά τα άλλα έχουμε ένα πρόβλημα το brain drain, την διαρροή εγκεφάλων. Δεν επιθυμούμε οι ερευνητές μας να εγκαταλείπουν την Ευρώπη. Στον τομέα της έρευνας εργάστηκα επί τρεις δεκαετίες ολόκληρες Ομιλώ εκ πείρας λοιπόν και γνωρίζω το τι συμβαίνει. Οι δικοί μας ερευνητές είναι εξίσου καλοί όπως άλλοι ερευνητές και ελπίζω ότι σε αυτό το πεδίο θα μπορούσαμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και να σταματήσει πια αυτή η απορροή, η διαρροή εγκεφάλων, brain drain. Μιλάμε συχνά για την αριστεία, αλλά αναφέροντας την αριστεία είναι πολύ σημαντικό τα δικά μας ερευνητικά ιδρύματα να τα υποστηρίξουμε και να τα ενδυναμώσουμε. Χρειαζόμαστε μια, ένα καλό συμβιβασμό λοιπόν και αυτό θα έπρεπε να μας κινεί. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. καλώ ήρθατε, κυρία Επίτροπε. Νομίζω ότι θα είμαστε στρατηγική εταίροι για τους επόμενους μήνες, αν θέλετε κι εσείς να κερδίσουμε τη μάχη μεγιστοποίηση των κονδυλίων έρευνα για την Ευρώπη. Νομίζω ότι είναι κοινό το συμφέρον μας. Είμαι συγγήτρια για το τμήμα του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου που ασχολείται με αυτά. Έχω λοιπόν τις ερωτήσεις ως εξή. Πώς βλέπετε ότι μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε τα δημοσιονομικά μέσα και να πείσουμε το Συμβούλιο και ιδίω μιλώντας για χώρες όπως τη δική μου που ε, ενδιαφέρονται μόνο για το Ταμείο Συνοχής. Πώς μπορούμε να αλλάξουμε τη γνώμη τους, πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την αριστεία και όχι μόνο διευκολύνσεις συνδέοντας την Ευρώπη για την ψηφιακή διασύνδεση και να διασυνδεθούν και τα ερευνητικά κέντρα. Ή τα αφήνετε τα κέντρα αριστείας για την πολιτική συνοχή μόνο ή πρέπει να σχεδιάσουμε συνεργασία και για αυτά. Ένα μέρος των χωρών μελών του Συμβουλίου νομίζομαι ότι θα θέλουν να το κάνουν αυτό. Και αν θέλουμε βέβαια και όπως θέλουν και ορισμένες χώρες να σταματήσουν την διαρροή εγκεφάλων από, από την ε, Ευρώπη. Το άλλο θέμα είναι ότι θέλουμε να διασώσουμε το ίτερ, το ΚΟΣΜΕ και άλλα προγράμματα. Και κυρίως βέβαια θέλουμε να διασώσουμε πρωτίστως τον ορίζοντα 2020. Δεν δεχόμαστε όμως να γίνουν περικοπές στο κεφάλαιο 5. Όταν μιλούμε για ερευνητικά προγράμματα, χρειαζόμαστε την τα διοικητικά κονδύλια. Χρειαζόμαστε και το προσωπικό τη Κομισιόν. Δεν μπορούμε λοιπόν να χάσουμε χρήματα ούτε εκεί. Πώς λοιπόν μπορούμε να συνασπιστούμε, να συμμαχίσουμε ώστε να εργαστούμε έτσι για υπέρ της Ευρώπης. Τελευταίος παρεμβαίνων για μισό λεπτό κυρία Τικάου, για μισό λεπτό παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πέραν της έρευνας για την ανάπτυξη τεχνολογίας στον πυρηνικό τομέα, τονίζω ότι χρειάζεται συνεργασία σε διεθνές επίπεδο και για την πυρηνική ασφάλεια, διότι τα ε, πυρηνική σταθμή μας είναι ήδη ηλικία πολλών δεκαετιών και εκτός αυτού παράγουν και πολλά κατάλοιπα. Έτσι λοιπόν πρέπει να συνεργαστούμε και στον τομέα της ασφάλειας των πυρηνικών σταθμών. Τελειώνοντας ο κύριος Σοντή, μάλλον τελευταίος ο κύριος Σοντή. Ευχαριστώ. Η ανησυχία σήμερα των χωρών και των λαών είναι η ανάπτυξη. Ακούμε συχνά ότι η ανάπτυξη θα προκύψει από την έρευνα και την καινοτομία. Μήπως κατάλαβα ότι θα ρηχθεί ιδιαίτερο βάρος στη διεθνή συνεργασία μήπως πρέπει να στοχεύσουμε περισσότερο σε ανάπτυξη των επιχειρήσεών μας. Τελευταία ερώτηση. Μιλήσαμε πολύ για την πρόσβαση. Ανοίγουμε τα πάντα. Ωστόσο θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε τα αποτελέσματα της δημόσια χρηματοδοτούμενης έρευνάς μας υπέρ των επιχειρήσεών μας και επομένως με την προστασία των ευρεσιτεχνιών. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ για τις παρεμβάσεις σας και δίνω το λόγο στην κυρία Επίτροπο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ όλους τους συναδέφους. Νομίζω ένας από τους συναδέφους πρότεινε και είπε ότι ήμουνα εδώ με τον στρατηγικό μου εταίρο. Πράγματι, στη μάχη για τον προϋπολογισμό που έχουμε μπροστά μας. Είναι σαφές αυτό. Και δεν θα έπρεπε να παρεκκλίνουμε όσον αφορά τη διεθνή διάσταση. Βρισκόμαστε στον αγώνα της ζωής μας για την επιβίωση. Ακούμε από την Κορεπέρ, αυτά τα οποία ακούμε δεν μας, δεν μας γεμίζουν χαρά δεν είναι χαρμόσυνα μαντάτα. Υπάρχει μεγάλη μάχη μεταξύ ΚΑΠ και πολιτική συνοχή, μεταξύ κοινή αγροτική πολιτική και κονδυλίων για την πολιτική συνοχή. Εκείνοι που πρέπει να είναι προπομπή και πρωτοπόροι για τις επενδύσεις όσον αφορά την έρευνα και την ε, ανάπτυξη, όταν καταλήγουμε στο τέλος στα, στα παζάρια μεταξύ των δύο μεγάλων αυτών τομέων, ίσως ε, το εξυλαστήριο θύμα, ε, το θύμα που θα θυσιαζόταν θα μπορούσε να είναι η έρευνα και η ανάπτυξη. Δεν πρέπει να γίνει αυτό. Πρέπει να ενθαρρύνουμε τους ομολόγους και εταίρους μας, είτε είναι ερευνητές, είτε είναι επιχειρήσεις, θεσμικά ιδρύματα, να μπορέσουν να προαγάγουν το θέμα στα κράτη-μέλη και να επεξηγήσουν ότι αυτή είναι η πολιτική του μέλλοντος. Αυτή είναι η πολιτική που θα δώσει ανταγωνιστικότητα στις οικονομίες μας. Θα βοηθήσει τις οικονομίες μας να αναπτυχθούν και θα παράσχει θέσεις εργασίας και απασχόληση. Αυτά θέλω να πω μόνο όλοι γνωρίζω εργάζεστε για να υποστηριχθούν αυτοί οι στόχοι και να τα καταφέρουμε. Πρώτα απ' όλα τώρα για τη στοχοθετημένη συνεργασία και τις δράσεις. Θα υπάρξουν τέτοιες στοχοθετημένες δράσεις για τη συνεργασία όπου εμείς υπεύθυνοι για την πολιτική εκ προημίου θα αποφασίζουμε και τα παιδεία και τους εταίρους σε αυτή τη συνεργασία. Παράδειγμα, στον τομέα της ενέργειας θα ζητήσουμε συμβουλές φυσικά από τη Γενική Διεύθυνση για τα θέματα ενέργειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιο πριν σίγουρα για να θεσπίσουμε και να θεσμοθετήσουμε ποιοι τομεί στον τομέα της ενέργειας απαιτούν διευρυμένη διεθνή συνεργασία και θα καθορίσουμε τις χώρες που θα εμπλέκονται σε αυτή τη διεργασία που πρέπει να εντοπιστούν και να ταυτοποιηθούν. Δεν πρέπει να το κάνουμε εμείς ξεχωριστά αυτό για κάθε ένα από τους τομείς πολιτικών που ακολουθούμε. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα συνεργαστούμε με την αρμόδια Γενική Διεύθυνση που θα έχει συγκεκριμένε ευθύνε για ένα συγκεκριμένο πεδίο πολιτική. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι το πρόγραμμα έρευνα, το 7ο πρόγραμμα έρευνα και ανάπτυξη και ορίζοντα 2020 είναι ανοιχτά προγράμματα. Εδώ έχουμε και το θέμα των ε, όσων συμμετέχουν ε, στο ύψο του 5% σε αυτό το πρόγραμμα. Όμω πρέπει πολύ περισσότερα να κάνουμε ώστε να είναι πιο ευδιάκριτα όλα τα στοιχεία και οι πρωτοβουλίε. υπό το 7ο πρόγραμμα δράσης για την έρευνα και την ανάπτυξη και ο ορίζοντας 2020 να είναι ανοιχτή στα πλαίσια του για τον ιδιωτικό τομέα, τον κρατικό τομέα, του ερευνητέ, του επιστήμονε από όλες τις χώρες παγκόσμια. Είναι σημαντικό να το υπογραμμίσουμε αυτό, παρότι πολλοί από μας εδώ γνωρίζουν σήμερα ότι αυτό συμβαίνει και είναι δεδομένο. Για τη συγκεκριμένη αυτή ε, διεθνή συνεργασία και για τις ε, διαδικασίες που θα ακολουθηθούν με τις χώρες που έχουν συμφωνίες για την έρευνα και την ανάπτυξη με την ΕΕ. Υπό το 7ο πλαίσιο ο μονάδες και όργανα από όλε τις χώρες ε, ανάλογα με το ΑΕΠ ε, που έχουν χαμηλό, μεσαίο, ανώτερο ε, μπορούν να είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση, αυτόματη χρηματοδότηση. Και όπως λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κριτήρια για την θέσπιση, την κατάρτιση του, καταλο... του καταλόγου για την αυτόματη αυτή έγκριση χρηματοδότησης θα αναθεωρηθούν για τον ορίζοντα 2020 με πρόσθετα κριτήρια σε σχέση με το συνολικό συνολικό ΑΕΠ, αποκλείοντας ε, από χώρε που το ΑΕΠ του θα βρίσκεται πάνω από ένα συγκεκριμένο κατόφλι. Και αυτό αφορά τις χώρες εκείνες, ιδιαίτερα τις BRICS, που έχουν καθορίσει την, έχουν ε, θεσμοθετήσει την αναγκαία κριτική κρίσιμη μάζα που χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση για τέτοιου είδους δράσεις. Εξίσου για τη χρηματοδότηση εταίρων από τέτοιες χώρες ε, που θα μπορεί να διασφαλίζεται κατ' εξαίρεση υπό εξαιρετικές περιπτώσεις. Όλοι θα αξιολογούνται σε διετή, αναδιετή περίοδο με ανεξάρτητους ε, ε, αναλυτές και αξιολογητές. Είναι σημαντικό όταν θέτουμε στόχους με ε, οδικούς χάρτες να εξετάζουμε και να βλέπουμε, να διασφαλίζεται ότι αυτά τα οποία υποσχεθήκαμε θα επιτυγχάναμε, πράγματι θα επιτυγχάνονται για το ε, FP7 η αυτόματη χρηματοδότηση περιορίστηκε στις χώρες που δεν είναι υψηλού εισοδήματος, όπως είπα και για τα κριτήρια της Παγκόσμιας Τράπεζας πιο πριν, θα έχουμε φορείς που κατ' εξαίρεση θα μπορούν να χρηματοδοτούνται. Για παράδειγμα, όταν θα υπάρχει μια αμοιβαία συμφωνία, για παράδειγμα, όσον αφορά τις ίπα π.χ ή όπου είναι σαφές ότι η συνεισφορά του εταίρου της τρίτης χώρας αυτής θα είναι θεμελιώδους σημασία για να μπορέσει να στεφτεί με επιτυχία η μετεξέλιξη και η ολοκλήρωση ενός προγράμματος. Όλα αυτά σε σχέση με το πρόγραμμα του Ορίζοντα 2020 με την εξαίρεση ότι η αυτόματη χρηματοδότηση θα περιορίζεται όταν μια χώρα έχει υπερβολικά μεγάλο ΑΕΠ ακόμα και αν μια τέτοια χώρα δεν ε, έχει κατηγοριοποιηθεί ως χώρα ειδικά υψηλού εισοδήματος. Όσον αφορά τώρα για παράδειγμα τη Γεωργία. Απογοητεύτηκα που άκουσα ότι κάποιο ανέφερε ότι δεν υπήρχε καμία λέει αναφορά στη Γεωργία στον ορίζοντα 2020 στη στρατηγική μα. Παρέμβαση χωρί μικρόφωνο. Πώ είπατε, πολιτισμό. Permaculture. Πρέπει να μάθω τι είναι τα θέματα permaculture. Και σε σχέση με την γεωργία γενικότερα υπάρχει τώρα μια πιο στενή ε, εμπλοκή σε σχέση με τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και την Γενική Διεύθυνση Καινοτομίας και Έρευνας. Και προφανώς η αηφορία, η αηφόρος γεωργία είναι μία από τις παγκόσμιες ε, προκλήσεις. Ένα από, ε, ένας από τους έξι άξονες μέσα στο πρόγραμμα της στρατηγικής ορίζοντας 2020. Όπως είπατε είναι ένας αναπτυσσόμενος τομέας. Πολλές συναλλαγές μπορούν να γίνουν ε, και σε συνεργασία με διεθνεί διεθνείς εταίρους και να συνεργαστούμε με αυτούς τους διεθνείς εταίρους για την ανάπτυξη στρατηγικών υποδομές και υποδομές σε σχέση με την έρευνα είναι ευρύτερες και απαιτούν συνεργασία και υποστήριξη από αρκετές χώρες. Και όπως αναφερθήκατε στο ITER ως παράδειγμα, ένα άλλο παράδειγμα θα ήταν το CERN στην Ελβετία με την ε, ταυτοποίηση των ε, όσων πρέπει να γίνουν θα έχουμε έναν οδικό χάρτη για τις έρευνες και την χρηματοδότηση των υποδομών για την έρευνα την ΕΕ. Αυτό υπογραμμίζει πάντα την ανάγκη συνεργασίας, της πτυχής της συνεργασίας θα βασιζόμαστε πάντα στην πείρα που έχουμε συλλέξει διασυνοριακά σε τέτοιου είδους δράσεις συνεργασίας και θα λάβουμε φυσικά υπόψη το έργο που έχει επιτευχθεί από τους υψηλόβαθμους αξιωματούχους για τις υποδομές που θεσπίστηκε από την ομάδα των οκτώ των Υπουργών δηλαδή ε, για ε, τα θέματα επιστημών. Αυτό όσον αφορά το πλαίσιο της παγκοσμιοποιημένης έρευνας και τις υποδομές. Θα έλεγα πολλοί πάμπολοι αναφέρθηκαν στην ανάγκη του να υπάρξει η εμπλοκή και συμμετοχή της βιομηχανίας, των βιομηχανικών κύκλων και να είναι πιο εύκολο για τις μικρότερες ερευνητικές μονάδες ε, ε όσον αφορά την έρευνα να έχουν πρόσβαση σε ένα πολύ λιγότερο ε, με μικρότερη γραφειοκρατική επιβάρυνση πλαίσιο από ό,τι μέχρι σήμερα Γνωρίζετε, Κρόλεϊ, Ευρωβουλευτά, μία από τις κυριότερες προκλήσεις στην ανάπτυξη του ορίζοντα 2020 ήταν η ριζοσπαστική, ρηξικέλευτη απλούστευση. Και θέλω να τονίσω και πάλι πόσο εκτιμώ το έργο που έχει επιτευχθεί από αυτήν την Κοινοβουλευτική Επιτροπή, εμένοντας και επιμένοντας τον ορίζοντα 2020 ότι το κυριότερο στοιχείο, ο στόχος, πρέπει να είναι αυτή η εκβάθρον απλούστευση, εξαπλούστευση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτή η απλούστευση θα οδηγήσει σε μια κατάσταση, άσχετα από το πόσο μικρή μπορεί να είναι η εταιρεία σας το μέσο, το, ε, ο θεσμός τον οποίο υπηρετείτε να γνωρίζετε ποιοι κανόνες και κανονισμοί θα εφαρμόζονται και θα ερμηνεύονται ενιαία και θα υλοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση με μία θηρίδα που θα είναι αρμόδια με σεβασμό από όλους και ευθυγράμμιση σε όλες αυτές τις προδιαγραφές και ιδιαίτερα όσον αφορά και τις προδιαγραφές του χρηματοοικονομικού κανονισμού όλα αυτά ε, δουλεύουν ώστε να μπορούν, θα ε, ε, συνεργάζονται ώστε να μπορούν να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες όλων και των μικρών. Και είναι ένα θέμα τεράστια σημασία αυτό για τους Ευρωπαίους ερευνητές και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Προφανώς είναι ένα θέμα το οποίο έχει τα μέγιστα συνειδητοποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχω πολύ στενά συνεργαστεί με τον Επίτροπο κύριο Μπαρνιέ για ένα νέο καταστατικό και καθεστώς για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και των προϊόντων των δημιουργών. Έχετε δει βήματα που έχει κάνει ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προτίθεται να κάνει και άλλα στο μέλλον. Θα ακολουθήσουν και άλλα βήματα. Αυτά είναι κυριότερα μελήματά μας, τα οποία πράγματι θέλουμε να επιτευχθούν. Και Θέλουμε να έχουμε ένα σύστημα που θα προστατεύει και θα υποστηρίζει τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών εδώ στην Ευρώπη. Φυσικά έχετε δίκιο όταν λέτε ότι είδαμε έρευνα που επετέφθη στην Ευρώπη να την εκμεταλλεύονται εμπορικά αλλού σε άλλες υπήρους και για τις διάφορες τεχνολογίες που αναφέρατε. Αυτό, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε η πρωτοβουλία καινοτομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να ξεπεράσουμε τέτοια προβλήματα και αντικσοότητες. Στο μέτρο του εφικτού να διασφαλίσουμε ότι όταν παράγουμε εμεί έρευνα εδώ στην Ευρώπη να, μπορεί να, να μπορούμε να την εκμεταλλευόμαστε εμείς εδώ στην Ευρώπη εμπορικά για την ταχύτερη διαδικασία ε, τυποποιημένων διατάξεων που θα πρέπει να ακολουθούνται ώστε να μπορούμε να προχωρούμε από ένα κράτος να μπορούμε να περνάμε σε άλλο πανενοσιακά θέματα όπως προμήθειες ε, ε, όπως το SPR Facility όπως έγινε και στη ΣΥΠΑ εξάλλου για όλα αυτά. Όλα αυτά είναι στοιχεία πολυσχηδή που θα βοηθήσουν και θα συνεισφέρουν να διασφαλίσουμε ότι αυτά τα οποία παράγουμε και δημιουργούμε στην Ευρώπη θα μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε εκμεταλλευόμαστε εμπορικά στην Ευρώπη όπου είναι αυτό εφικτό και δυνατό να δω μια στιγμή. Μάλιστα, νομίζω ότι προσπάθησα στο μέτρο του εφικτού, το καταδύναμη πρόεδρε, να απαντήσω στι παρεμβάσει και τα σχόλια των μελών. Για άλλη μια φορά θα ήθελα να εκφράσω τι ευχαριστίε μου που μου επιτρέψατε να παραστώ εδώ σε αυτή τη συζήτηση και να είμαι παρούσα σήμερα εδώ. Δεν υπάρχουν σύνορα σε όλα αυτά. Συνεργαστήκαμε διεθνώ με μεγάλη επιτυχία στο παρελθόν και θέλω να διασφαλίσω προσωπικά ότι η στρατηγική του ορίζοντα 2020 ε, θα είναι εξίσου ανοιχτή όπω και τα προγράμματα πλαίσια για την έρευνα και την ανάπτυξη μέχρι σήμερα. Προσβλέπω σε αυτό, ιδιαίτερα και δεδομένη τη δημοσιονομική αντιπαράθεση που βρίσκεται υπό εξέλιξη. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστώ εκ μέρου ε, όλων των συναδέλφων της Επιτροπής μας. Σας ευχόμαστε καλή δουλειά και ε, θα τα ξαναπούμε στο επανειδή. Πάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα ε, της σημερινής μας συνεδρίασης. Το επόμενο θέμα αφορά στις δυνατότητες που έχουμε αυτή τη στιγμή για τις ανανόσιμες πηγές ενέργειας ε, στην εσωτερική αγορά ενέργειας. Έχουμε λοιπόν εδώ και την παρουσία της Άρτε, της ε, τηλεοπτικής ομάδας που κάνει ένα ντοκιμαντέρ για την ενέργεια. Και δίνω μέσα στο λόγο ε, στον εισηγητή σας, τον Αλφα κύριο Ρόιλ. Παρακαλώ. Μισό λεπτό, αν έχετε καλωσία να περιμένετε να βγουν όλοι όσοι δεν ενδιαφέρονται. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, Σήμερα έχουμε την πρώτη συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων για το θέμα αυτό. Είναι ένα θέμα το οποίο αναμφισβήτητα είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για το μέλλον της, ε, του ενεργειακού εφοδιασμού. Να πω λοιπόν ευθύ εξ αρχής ότι υπάρχει ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία κατά την άποψή μου αποτελεί μια καλή περιγραφή της κατάστασης που επικρατεί στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ευρώπη. Φύγει αυτή η ανακοίνωση πολλά και σημαντικά θέματα. Και στο θέμα αυτό δεν ξεκινάμε από το μηδέν, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν χρειάζεται δηλαδή να συντάσουμε μακροσκελή έγγραφα για να αποδείξουμε ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι καθοριστική σημασία για τον ενεργειακό ανεφοδιασμό του μέλλοντος. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο και θα αναφέρω σήμερα κάποιες απόψεις γιατί θέλω να γνωρίζω τι πιστεύουν οι συνάδελφοι. Βέβαια την έκθεση δεν την έχω ακόμα στην τάξη, στην τελική της μορφή και θα λάβω υπόψη με αυτά που θα πούν οι συνάδελφοι. Καταρχήν, είναι σαφές ότι οι ανανεώσιμες πηγές ε, ε, διαδίδονται πολύ περισσότερο από ό,τι περιμέναμε. Και ενδεικτικά θα αναφέρω οι εγκατεστημένες μονάδες το 2007 σχεδόν δεκαπλασιάστηκαν. Και παρόλα αυτά βλέπουμε ότι πάνω από δύο τρίτα επιδοτούνται. Δηλαδή υπάρχουν αυτοί οι αριθμοί που είναι λίγο περίεργοι, προκαλούν ερωτηματικά και νομίζω ότι πρέπει λιγάκι να τους δούμε αυτούς τους αριθμούς. Γιατί αν υπάρχει ή αν θέλουμε μεγαλύτερο ποσοστό ανανεώσιμων πηγών, υπάρχουν κάποια ερωτήματα που πρέπει καταρχήν να τεθούν, κατά δεύτερον να απαντηθούν και Βεβαίως δεν είναι τίποτα το, γεγον, το καινούριο ότι η ε, ασφάλεια αναφοδιασμού, η βιωσιμότητα, αυτά είναι σημαντικά στοιχεία. Ξεκινάω λοιπόν με ένα θέμα και κάποιες ερωτήσεις. Πιστεύω, ένα από τα βασικά στοιχεία αυτή τη στιγμή και όχι όταν ξεκινήσαμε, αλλά τώρα. Καθοριστική σημασία είναι το θέμα του κόστους. Κόστος λοιπόν των ανανεώσιμων πηγών. Γιατί μέχρι τώρα στην Ευρώπη, εκεί όπου υπάρχουν εκτεταμένες τέτοιες δομές, είναι πολύ δαπανηρές. Καταρχήν για την επιδότηση, αυτό ε, μετακυλίεται στους ε, καταναλωτές και φτάνουμε σε ένα σημείο όπου πολλές φορές οι πελάτες δεν επιθυμούν τις ανώσιμες πηγές. Λένε, μα δεν μπορούμε πια να αντιμετωπίσουμε αυτό το κόστος. Δεύτερον, η υποδομή. Εδώ μιλάμε για υποδομές που όμως δεν είναι αποκεντρωμένες, δεν είναι προσαρμοσμένες στην αποκέντρωση. Και τέλος έχουμε τα αποθέματα τα οποία είναι σημαντικά για τις συμβατές ε, μορφές ενέργειας. Η συμβατή ενέργεια δεν ε, εξαφανίζεται, απλά υπάρχει παράλληλα στη Γερμανία. 12 δις ευρώ δίδονται σε τήσια βάση με τη μορφή επιδότησης. Και εντωμεταξύ Μιλάμε για τεράστια ποσά, ε, το κόστος της ενέργειας αυξάνεται συνεχώς, άρα δηλαδή αυτό είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί. Πώς μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτά τα προβλήματα. Βεβαίως ισχύει και το αντίθετο, ότι ένα τμήμα των χρημάτων στην Ευρώπη δεν είναι ότι δαπανάτε, δημιουργούνται νέε θέσει εργασία. Αυτό είναι πολύ καλό. Στη δική μου τουλάχιστον την πατρίδα, ε, πολλέ ε, μονάδε ηλιακή ενέργεια δεν παράγονται πλέον στην Γερμανία, αλλά στην Κίνα. Που σημαίνει ότι με τα λεφτά του Γερμανού φορολογούμενου ε, επιδοτούμε την κινέζικη βιομηχανία. Και καταλαβαίνετε, εδώ δεν μπορεί να συνεχιστεί. Πρέπει κανεί να έχει το θάρρο να δει να πει να δούμε τώρα τι θα κάνουμε. Όσον αφορά τώρα τις υποδομές, ε, χρειαζόμαστε τελείως διαφορετικές υποδομές από ό,τι μέχρι τώρα, διότι ε, τα συστήματα εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες, δεν είναι μόνιμες εγκαταστάσεις. Αναφέρθηκε ότι το 80% όλων των προβλημάτων στις, ε, στον ενεργειακό ανεφοδιασμό είναι σε άμεση έμεση σχέση με τις ανανεώσιμες πηγές. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν είναι καλές αυτές, αλλά είναι ένα πρόβλημα και το πρόβλημα πρέπει κανείς καταρχήν να το ονοματίσει για να βρει μετά τη λύση. Άρα δηλαδή χρειαζόμαστε νέες υποδομές, νέα δίκτυα, χρειαζόμαστε τη δυνατότητα αποθήκευσης. Αυτό πάλι κοστίζει χρήματα. Τρίτο σημείο και θα αναφερθώ ε, στον έλεγχο γενικότερα της εργαλειοθήκης ε, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά πολλοί λένε δικαίως ότι οι τιμές των εκπομπών είναι πολύ χαμηλές. Αυτό όμως έχει άμεση σχέση με την οικονομική κατάσταση και έχει και άμεση σχέση με το ότι χρειαζόμαστε τόσο μεγάλη επέκταση των ανανεώσιμων πηγών και αν αυτές αντικαταστήσουν τις συμβατές, ε, ε, στην περίπτωση αυτή βέβαια και είναι πιο ευνοϊκές, ε, είναι πιο φτηνές αυτές οι μορφές ε, ενέργειας. Άρα δηλαδή τι θα γίνει. Ε, θα πέσουν οι τιμές στην ανταλλαγή των ποσοστώσεων εκπομπών. Αυτό που ενδιαφέρει είναι το εξής. Μπορούμε μακροπρόθεσμα να επιδιώκουμε τόσους πολλούς και παράλληλους στόχους στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής. Μήπως θα ήταν πιο έξυπνο να προχωρήσουμε στοχευμένα, γιατί ναι μεν καλό το να υπάρχουν ε, πολλοί και παράλληλοι στόχοι, ε, καθησυχάζει την κοινή γνώμη το να παρουσιάζονται καινούργια στοιχεία, όμως αυτό δεν ξέρω αν είναι αποτελεσματικό. Μπορεί πολλές φορές να δημιουργεί και πρόβλημα. Και το τελευταίο που θέλω να αναφέρω είναι το εξή. Έχει σχέση με αυτό που ανέφερα, τις επιδοτήσεις. Οι επιδοτήσεις δεν είναι βιώσιμες. Είναι πάρα πολύ δαπανηρό το όλο σύστημα και οι επιδοτήσεις στις ανώσιμες πηγές δημιουργούν και ανισότητες στην Ευρώπη. Για να ολοκληρωθεί λοιπόν η κοινή αγορά θα πρέπει να μην υπάρχει αυτό το μοσαϊκό, το εμβαλωματικό μοντέλο από ε, διάφορες ε, εκπομπές ε, και ανταλλαγή εκπομπών. Αν κάποιος ας πούμε αποφασίσει να επενδύσει στη Βόρειο Ελλάδα και όχι στην Ελλάδα, την ηλιακή ενέργεια, πρέπει κανεί να διερωτηθεί, μα μήπω εδώ πρόκειται για διασπάθηση χρήματο. Βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου θα πρέπει να σκεπτόμαστε πώ μπορούμε να επενδύσουμε σωστά τα δημόσια κονδύλια. Είναι δυνατόν στη Βόρεια Γερμανία να επενδύονται τεράστια κονδύλια, ενώ στην Ελλάδα οι ανανόσμες πηγές είναι πολύ πιο φτηνές και μάλιστα πολύ πιο αποτελεσματικές, γιατί είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα υπάρχει μεγαλύτερη ηλιοφάνεια. Ε, η Επίτροπος το επισήμανε το θέμα αυτό. Επίσης, η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της, και αυτό για μένα είναι καθοριστική σημασία, ε, τοποθετήθηκε και στην πολιτική συζήτηση. Κατά πόσον δηλαδή επιθυμούμε να έχουμε στενότερο και ουσιαστικότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο στην όλη συζήτηση. Μπορούμε να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο ε, την ενεργειακή πολιτική όπως το κάνουμε, δηλαδή κάθε χώρα να κάνει ό,τι θέλει ή μήπω έχει φτάσει η στιγμή όπου θα πρέπει να προσπαθήσουμε τις ανανεώσιμες πηγές να τις ε, προάγουμε περισσότερο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δηλαδή να εξευρωπαίσουμε τα ε, συστήματα. Αυτό βέβαια δεν γίνεται εν μια νυχτή και γνωρίζω και την πολιτική πίεση που ασκείται στα κράτη-μέλη. Όμως το να επιδείξει κανείς ρεαλισμό δεν βλάπτει μικρότερη κατάτμιση, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, μεγαλύτερη διάδοση, μεγαλύτερη αξιοπιστία. Ε, αυτή θα ήθελα να είναι η ανακοίνωσή μας. Περίπου. Όχι να είναι ένα μακροσκελές έγγραφο που θα παραλαμβάνουμε τα ίδια και τα ίδια, αλλά να εστιάσουμε την προσοχή μας στα σημεία εκείνα που ενδεχομένως θα πρέπει να αντιπαρατεθούμε με το Συμβούλιο και όπου θα προχωρήσουμε μόνο αν κατορθώσουμε να απαντηθούν τα θέματα αυτά τώρα. Πολύ καλύτερα τώρα από ό,τι πριν από τρία-τέσσερα χρόνια όταν ξεκινήσαμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και με μεγάλη μου χαρά και ανυπομονησία περιμένω να δω τι θα προσθέσετε έτσι ώστε να καταλήξουμε σε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία, λέει η Πρόεδρος. Ε, ξεκινάει λοιπόν η συζήτηση και έχουμε στη διάθεσή μας 45 ε, λεπτά. Άρα δηλαδή ε, ξεκινώ δίνοντας το λόγο στον κύριο Λάγκε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καθώς επίσης και σας κύριε Ρόελ. Πέντε θέματα θέλω να θίξω που με συγκινούν ιδιαίτερα και ορισμένα βέβαια τίνουν να συμφωνήσουν και με αυτά που είπατε, κύριε Ρόιλ. Βλέπω και εγώ ότι επί της παρούσης στην πολιτική της ενέργειας έχουμε πράγματι ένα ευρύτατο φάσμα το οποίο επιδιώκουμε να υλοποιήσουμε και χρειάζεται πράγματι να δούμε που μπορούμε ίσως να συγκεντρώσουμε καλύτερα τις προσπάθειές μας και τις δραστηριότητές μας. Όλη αυτή η υπόθεση για την ανταλλαγή, ε, με την εμπορία των ε, εκπομπών νομίζω ότι προσανατολίζει. Όπως ε, προβλέπεται και στο έγγραφο για το 2020 πρόκειται για ανανεώσιμες ενέργειες και για αποδοτικότητα της χρήσης της ενέργειας. Κατά τη γνώμη μου χρειάζεται μια συνεπή συνεκτική πολιτική η οποία να λαμβάνει υπόψη και τις δύο αυτές παράλληλες τροχές μέχρι το 2020 έτσι ώστε να μειωθεί σιγά σιγά η εξάρτηση από τις ορυκτές πηγές καυσίμων. Γι' αυτό λοιπόν εδώ συμφωνώ ότι πρέπει να ρίξουμε περισσότερο το βάρος. Μιλώντας τώρα για τις ανανεώσιμες ενέργειες, αυτά τα πέντε θέματα που σας ανέφερα προηγουμένως είναι τα εξή. Έχουμε το δεσμευτικό στόχο μέχρι το 2020 ε, του ποσοστού 20% της συνολικής ε, ε, χρησιμοποιούμενης ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Θα το επιτύχουμε, έστω και αν με διαφορετικά ποσοστά αναχώρα, αλλά στο σύνολο θα το επιτύχουμε. Το ερώτημα που θέτω εγώ είναι μετά τι γίνεται θα πάμε έτσι μέχρι το 2020 και έχουμε και τον οδικό χάρτη ενέργεια 2050 ή θα βάλουμε κάποια ενδιάμεσα στάδια ώστε να καταστεί σαφές προς τα πού επιθυμούμε να κινηθούμε και ποια είναι τα πολιτικά εκείνα μέτρα που θα πρέπει να λάβουμε. Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο. Δηλαδή πώς, τι μορφή θα λάβει αυτό το χρονοδιάγραμμα. Και ύστερα κύριε Ρόιλ πράγματι το ζήτημα των ενισχύσεων, είναι σαφές, ίσως όχι όλες οι ανανεώσιμες ενέργειες, να διατίθενται σε τιμές αγοράς ή πάντως να παράγονται σε τιμές αγοράς. Θα χρειάζεται λοιπόν, επειδή δεν μπορούν να παράγονται σε τιμές αγοράς, και κάποιες ενισχύσεις. Όμως ούτε εδώ μπορεί να είναι ένα patchwork όπως λένε στα αγγλικά. Δηλαδή τα διαφορετικά συστήματα ενισχύσεων έχουν αποδώσει διαφορετικά αποτελέσματα από αυτό το σύστημα το οποίο διοχετεύουν ιδιώτες ρεύμα που παράγουν στο κεντρικό δίκτυο μέχρι άλλα συστήματα, μέχρι το μοντέλο των ποσοστώσεων και ούτω καθεξής με πολύ διαφορετικά αποτελέσματα. Αφετέρου, κάτι το οποίο έχει προκληθεί και ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση, σημαντικές τρευλώσεις του ανταγωνισμού σε ό,τι αφορά τις τιμές. Και τα δύο αυτά επιχειρήματα οδηγούν στο να σκεφτούμε ότι χρειάζεται περισσότερη ευρωπαϊκοποίηση του συστήματος ενισχύσεων, ώστε να φύγει από τη μέση και αυτό το κατακαιρματισμένο patchwork, αν δούμε τις ορισμένε περιφέρειες της Ευρώπης, εκεί όπου υπάρχει ίσως πολύ δυνατός άνεμος, υπάρχουν λίγες ανεμονογεννήτριες. Και αφετέρου, η στρεβλώση του ανταγωνισμού επίσης είναι σημαντικό να εξαλειφθούν. Και επίσης το τρίτο θέμα, δυστυχώς είναι ανοιχτό το μικρόφωνο τη Προέδρου η οποία ομιλεί. Τώρα το έκλεισαν, ευχαριστούμε πολύ. Είναι και αυτό πρέπει να είναι λοιπόν κοινό στόχος και χρειάζεται επομένω σημαντικότερη, περισσότερη κοινοτικοποίηση των πολιτικών. Άρα να σκεφτούμε επίσης με ποιον τρόπο θα εμπορευτούμε τις ανανεώσιμες ενέργειε και πώς θα διασφαλίσουμε τις επενδύσεις. Παράδειγμα Ελλάδα. Εν ώψη της κατάστασης που διαμορφώνεται εκεί, ορισμένοι δηλαδή σκέπτονται ότι η Ελλάδα θα πρέπει να εγκαταλείψει την Ευρωζώνη, ε, βέβαια αυτό δεν προσφέρει καμιά ασφάλεια στους επενδυτές. Τρίτο λοιπόν, κοινοτικοποίηση της πολιτικής εκμετάλλευσης των ανανεώσιμων ενεργειών, καθώς και σταθερή όρη για την εξέλιξη των ανανεώσιμων ενεργειών. Τέταρτο, πράγματι η πολιτική υποδομών που έχει άμεση σχέση. Στην ανακοίνωση λίγα λόγια περιλαμβάνει, αλλά το ζήτημα των ευφυών δικτύων, smart grids, είναι απόλυτα απαραίτητο να τεθεί και εδώ, διότι χρειαζόμαστε σαφώς και αποκεντρωμένες ε, ε, πυρήνες δημιουργίας της ενέργειας, παραγωγής της ενέργειας. Και εν τέλει οι ε, επενδύσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ ωραία. Ε, συνάδελφος Αλ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ εσάς ε, κύριε Ρόζ για αυτά τα οποία κάνατε. Είναι πολλές ε, προκλήσεις και πολλές ευκαιρίες που προσφέρονται όπως τίθεται και από την έκθεσή σας και για τα θέματα τα οποία πρέπει να προσέξουμε και να συζητήσουμε σε αυτή τη συζήτηση. Είναι σημαντικό πιστεύω να θυμόμαστε πάντα το γενικότερο πλαίσιο, γιατί χρειαζόμαστε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πρέπει να μειώσουμε τις εκπομπές άνθρακα στην ατμόσφαιρα και τα επιστημονικά τεκμήρια δείχνουν ότι αυτό είναι πολύ πιο κατεπήγον από ό,τι πιστεύαμε παλιότερα. Βλέπουμε ότι η εμπορία ρήπων αφεαυτής δεν λειτουργεί ως ε, ένας αποτελεσματικός κινητήριος μοχλός με κινητήρια μηχανή για όλα αυτά. Τι συμβαίνει στην πραγματικότητα επιτόπου. Τα ανανεώσιμα κάνουν την πολύ σημαντική βαριά δουλειά για την μείωση των εκπομπών άνθρακα. Η στρατηγική για τον ορίζοντα 2020 είναι κάτι το πολύ φιλόδοξο για την μείωση των εκπομπών ρήπων. Οι άλλες εναλλακτικέ επιλογές όμως χωλαίνουν κάπως. Δεν υπάρχει νέα πυρηνική συνιστόσα το κόστος συνολικά μετά την Φουκουσίμα είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικό και βλέπουμε ότι πολλά πράγματα ακολουθούν βραδύτα τους ρυθμούς και τα πιλωτικά προγράμματα ε, χωλένουν, έχουμε μεγάλη πορεία που πρέπει να καλύψουμε. Τα ανανεώσιμα λοιπόν είναι εκείνα από τα οποία εξαρτώμαστε για να καταφέρουμε να πετύχουμε αυτή τη σημαντική μείωση στην ατμόσφαιρα των εκπομπών άνθρακα όπως χρειάζεται και έχει νόημα και πραγματιστικά, ρεαλιστικά να τα δεχθούμε αυτά ως δεδομένα και να ακολουθήσουμε ε, μια πορεία για τα ανανεώσιμα μέχρι το 2030 αξιόπιστη και λειτουργική. Ιδιαίτερα είναι σημαντικό στοιχείο αυτό για τους πολίτες. Είναι πολύ σημαντικό να έχει εμπιστοσύνη σε αυτές τις συνιστώσεις και τις κατευθύνσεις οι βιομηχανίες. Τα ανανεώσιμα έχουν το ρόλο τους να διαδραματίσουν για να διεξέλθει η Ευρωπαϊκή Ένωση από την ύφεση. Τεράστιες ε, ευκαιρίες και πολλές θέσεις απασχόλησης μπορούν να δημιουργηθούν. Χίλιες θέσεις ε, εργασίας ε, αναγιγαβάτα ε, όσον αφορά την αιωλική ενέργεια και θα πρέπει να τα δούμε αυτά μέσα σε ένα πιο εξειδικευμένο πλαίσιο και για την εισαγωγή των κυψελών από την ε, ε, Κίνα για τα, ε, την δυνατότητα εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας, η εμπλοκή και δέσμευση από της Ευρώπης για τις ανανεώσιμες ενέργειες πρέπει να δώσει δυνατότητα να δοθούν κίνητρα στις ευρωπαϊκές βιομηχανίες για να είμαστε ανταγωνιστικοί για το θέμα του κόστους. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να μην συγχαίουμε τα πράγματα και δημιουργείται σύγχυση γιατί ε, εδώ έχουμε και τα, τους λογαριασμούς που αυξάνονται. Ο πρώην ε, υπεύθυνο για τα ενεργειακά θέματα στο ε, Ηνωμένο Βασίλειο έκανε αναλύσεις επ' αυτού και δύο τρίτα των ορυκτών καυσίμων, δύο τρίτα σε σχέση με τον λογαριασμό και την, την αύξηση των λογαριασμών οφείλονται στις αυξημένες τιμές των καυσίμων, ορυκτών καυσίμων ε, όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο που εισάγουμε. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά διότι αφορούν το ευρύτερο θέμα της ενεργειακής τροφοδότησης και της ενεργειακής ασφάλειας και της μεγαλύτερης εξάρτησης που έχουμε ως Ευρωπαίοι. Αν ε, παράγουμε εμείς οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι τις δικές μας, ε, ε, τα δικά μας ενεργειακά προϊόντα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τότε δεν θα εξαρτώμαστε σε τόσο μεγάλο βαθμό από ρηκτά καύσιμα και προϊόντα τα οποία εισάγουμε από άλλες χώρες. Και έτσι λοιπόν θα πρέπει να μπορέσουμε να δώσουμε συνέχεια. Υπάρχουν πολλές διεργασίες που βρίσκονται υπό εξέλιξη και που θα μας βοηθήσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό για να τα πετύχουμε και με υψηλό ακόμα ποσοστό ανανεώσιμο ή με ένα μείγμα ενέργειας. Θα πρέπει σε μια αγορά να μπορεί κανείς να μεταξύ αυτών και πρέπει να υπάρχει ε, διασύνδεση μεταξύ των χωρών για να λειτουργήσει μια τέτοια στρατηγική και κάτι παραπάνω ακόμα. Αν έχουμε καλές διασύνδεσεις μπορούν, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις μονάδες αποθήκευσης που θα είναι διαθέσιμες σε πολλές χώρες. Και τέλος θα ήθελα να πω ότι για το θέμα της διαμόρφωσης τιμολογίων και τιμών δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα ανανεώσιμα είναι μια σχετικά πολύ νέα τεχνολογία και για την μείωση των τιμών υπολογίζεται ότι τα ηλιακά πάνελ θα είναι βιώσιμα από κοστολόγηση κοστολόγησης τιμολογίων και διαμόρφωση τιμών από το 2020 και εφ' Ένα θέμα θέλω να αναφέρω ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αν πάμε υπερβολικά γοργά στην παραγωγή ανανεώσιμων και όχι με αηφορία τότε αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα. Και θα θέταμε, για παράδειγμα, μονομερώς ε, θα αναλαμβάναμε κάποιες πρωτοβουλίες ε, και δεν θα βλέπαμε τις ευκαιρίες ανάπτυξης ε, πανευρωπαϊκά. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες εναρμονισμού και μπορούμε μακροπρόθεσμα να τις εκμεταλλευτούμε. Πρέπει να είμαστε όμως συνετοί και προσεκτικοί, μια και είναι μια νέα βιομηχανία αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Τούρμες παρακαλώ. Vielen Dank. Ähm, Ευχαριστώ. Ο κ. Ρόιλ λέει ότι οι ανανεώσιμες ενέργειες είναι δαπανηρές, ότι θα σημειώσουν, θα είναι ανάγκη μάλλον τεράστιων επενδύσεων και λέει μετά να μην βάλουμε άλλου νέους στόχους και ταυτόχρονα εναρμόνιση, πιθανότατα δηλαδή ένα μοντέλο ποσοστώσεων για την Ευρώπη. Αυτό θέλετε, ποσοστώσεις για την Ευρώπη. Μα δεν έχω, δεν έχω τοποθετηθεί οριστικά, ούτε ξέρω τι μου λέτε. Εγώ επαναλαμβάνω αυτά που είπες, λέει ο κύριος Τόρμες. Καλά λοιπόν, για το κόστος τώρα. Ανεμογεννήτριες onshore είμαστε στα 5-6 cent στις ε, καλύτερες τοποθεσίες και τα κόστη αυτά μειώνονται κιόλας. για το PV και αυτό είναι μεγάλο θέμα στη Γερμανία. Ναι, τα έτη 2010 και 2011 είχαν ακουστεί τότε και κριτικές φωνές όταν χρησιμοποιούνται τόσο πολύ τα φωτοβολταϊκά πρέπει ε, να σημειωθεί ότι θα υπάρχει και βάρος πλέον από το παρελθόν. Και το λέω αυτό και για τη δική μου πολιτική ε, οικογένεια. Με ακούλπα επομένω είναι και δικό μα το φταίξιμο γιατί το δέχτηκαν τελικά οι δικοί μα, οι πράσινοι, αλλά και οι άλλε ε, και, τα άλλα κόμματα ε, τα προώθησαν πολύ τα φωτοβολταϊκά. Σήμερα βλέπουμε ότι τα φωτοβολταϊκά τα είχαμε με τότε και τα βάζαμε στις στέγες μας με 15 σέντ το κιλοβάτ, την κιλοβατόρα, κιλοβατόρα. Τώρα όμως για μεγάλες μονάδες στο νότο της Ευρώπης για τα φωτοβολταϊκά μπορούμε να φτιάξουμε με 9 ως 11 λεπτά του ευρώ την κιλοβατόρα. Αυτό είναι πραγματικά τεράστιο. Υπάρχει, ε, έγινε το μέγα αυτό ποιοτικό άλμα που χρειαζόμασταν. Εάν τώρα κάνουμε, ασκήσουμε μια ευφυή πολιτική ε, χρήσης φωτοβολταϊκών, μπορούμε να τα καταφέρουμε με κόστος που να ε, συμβαδίζει με τις νέες ε, εγκαταστάσεις. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε βέβαια το κόστος του ρεύματος από φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με τα παλαιά ε, με τις παλαιές εγκαταστάσεις καύσης άνθρακα ή πυρηνικές οι οποίες έχουν ήδη αποσβεστεί ως επενδύσεις. Χρειαζόμαστε λοιπόν διότι ένα νέο εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας είναι περίπου, η κιλοβατόρα κοστίζει 9 με 11 σεντ λεπτά του ευρώ. Όμως συνεπάγεται πολύ, βαρύτερες, πολύ κινδύνους και συνέπειες. Ο άνθρακας χωρίς το σύστημα CCS, συλλογής δηλαδή του, του, του καυσαερίου, του διοξιδίου του άνθρακα, δεν αντέχεται από το περιβάλλον. Άρα δεν είναι αλήθεια ότι η επέκταση των ε, ανανεώσιμων ενεργειών θα συνεπιφέρει τεράστιο κόστος. Για τις επενδύσεις τώρα και για τις επενδύσεις έχουμε φτάσει πλέον στην, ε, στο τέλος του πρώτου κύκλου. Και ε, δείτε ένα χάρτη της Γαλλίας της δεκαετίας του 70, το ίδιο και ένα χάρτη της Γερμανίας της δεκαετίας του 70, όπου υπήρχαν πολύ λίγες γραμμές υψηλής και άρχισαν να φτιάχνονται όταν άρχισε να λειτουργεί το γαλλικό και γερμανικό πρόγραμμα ε, Πυρηνική ενέργεια. Δηλαδή αυτό το rollout έγινε με τι πρώτε αυτέ επενδύσει στους πυρηνικούς σταθμού. και έγινε τότε μεγάλη επένδυση και στην υποδομή. Και γι' αυτό τα κόστη υποδομών, τα οποία μα αναμένουν ιστορικά, θα είναι στη τάξη μεγέθους εκείνων που έγιναν ήδη στι δεκαετίες 70 και 80, όταν επενδύαμε μαζικά σε ε, εργοστάσια ε, θερμικά και, δηλαδή άνθρακα, και πυρηνικά για την παραγωγή ενέργειας. Τώρα για τους στόχους. Φανταστείτε ότι σήμερα θα ήμασταν σε μια κατάσταση που να είχαμε μόνο το ETS, το σύστημα δηλαδή ανταλλαγή εμπορία ε, εκπομπών. Δεν θα είχε γίνει καθόλου ε, επένδυση σε ανανεώσιμες. Αυτό τα τρία πράγματα όμως, δηλαδή κλίμα, ανανεώσιμες και αποδοτικότητα τη ενέργειας έχουν το μέγα πλεονέκτημα ότι δίνουν στην οικονομία και στις τράπεζες που θα τα επενδύσουν αυτά τα πράγματα, θα, θα κληθούν να επενδύσουν αυτά τα πράγματα, μια ξεκάθαρη ορατότητα. Και εδώ όμως σημαίνεται μια μεγάλη αντίφαση. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι εναρμονίζω τα συστήματα ενισχύσεων, αλλά χωρίς στόχο. Δεν έχω στόχο ταυτόχρονα το μοντέλο ποσοστώσεων για την Ευρώπη ποιο θα είναι. Θα πρέπει να έχει ένα στόχο για την Ευρώπη 2030 και μετά να προχωρήσει σε ένα σύστημα ποσοστώσεων για να επιτευχθεί ο στόχος. Εδώ λείπει η λογική. Είτε υπάρχει στόχος για τις ανανόσιμες ενέργειες και τότε υπάρχει κάποια βάση για να συζητήσουμε ποιο θα είναι το σύστημα των ενισχύσεων. Ε, δεν μπορεί να γίνει αυτή η συζήτηση. Μια τελευταία λέξη για τη βιομηχανική πολιτική. Όπως είπε και ο Μπεντ Λάγκερ και προηγουμένω, το ότι σήμερα ερχόμαστε δεύτερη απέναντι στην Κίνα για την κατασκευή των λεγόμενων modules, τμήματων δηλαδή των ε, ε, εγκαταστάσεων, δεν είναι καλό. Και οι Κινέζοι κερδίζουν διότι δεν κερδοσκόπησαν οι τράπεζές τους για την κατασκευή αυτών των εγκαταστάσεων ε, ηλεκτρικής ενέργειας από, από τον ήλιο. Πρέπει λοιπόν να διαθέσουμε φθηνότερα κεφάλαια στις βιομηχανίες μας για να ανταγωνιστούμε τους Κινέζους. Και ο δεύτερος λόγος που η Κίνα παράγει φθηνότερα είναι ότι έχει πάρει τα καλύτερα γερμανικά, ελβετικά ή βορειοιταλικά μηχανήματα για την παραγωγή φωτοβολταϊκών βρίσκονται στην Κίνα. Οι πιο πρόσφατες εγκαταστάσεις, οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις έχουν γίνει στην Κίνα. Αν θέλουμε να ανταγωνιστούμε μαζί τους λοιπόν, πρέπει να διαθέσουμε φθηνότερα κεφάλαια και να δημιουργήσουμε αγορά. Τότε είμαι πεισμένος ότι θα τα καταφέρουμε. Η επόμενη γενιά εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών να φτιαχτεί στην Ευρώπη. Ο μέγας αγώνας σήμερα για τις εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών θα εξαρτηθεί από το ποιο είναι παραγωγικότερος και ποιο μπορεί να παράγει φθηνότερα. Και θέλω η Ευρώπη να αποδειχθεί ότι είναι αυτή. Βίδαλ Κουάρδας. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Υπενθύμιζε ο εισηγητής ότι πράγματι τις τελευταίες δεκαετίες η αύξηση των ε, ανανεώσιμο στην Ευρώπη ήταν κάτι εντυπωσιακό. Οι συνιστώσεις που οδήγησαν αυτή την εξέλιξη είναι αρκετά, είναι καλά γνωστή Η ανάπτυξη της ανάγκης να υπάρξει ενεργειακή ασφάλεια, ε, η αντιμετώπιση της απειλής των κλιματικών αλλαγών και οι προοπτικές όσον αφορά την αντικατάσταση των ε, ορυκτών καυσίμων με αυτά όλα κάναμε μια τεράστια προσπάθεια για να τα πετύχουμε και διπλασιάστηκαν από το 1995 μέχρι το 2010 ε, το ποσοστό. Τώρα είμαστε γύρω στο 10%. Μέχρι το 2020 θέλουμε να φτάσουμε το 20% στα ανανεώσιμα. Και η Ένωση και τα κράτη-μέλη εξίσου υποστηρίζουν στεναρά την ανάπτυξη των ανανεώσιμων μέσω των αναμφισβήτητων προτεραιμάτων που απορρέουν και όλοι συμφωνούμε ότι βρισκόμαστε σε μια μετάβαση προτύπου, μεταβατική περίοδο προτύπου, που θα εξαρτάται λιγότερο από τα ορυκτά καύσιμα, παρότι συνεχίζεται αυτή η συνιστόσα, αλλά λιγότερο θα εξαρτώμαστε από αυτά. Και θα δοθεί, λοιπόν, θα δοθεί το βάρος, όπως λέει ο δικός χάρτης μέχρι το 2005, σε αυτά. Αλλά προτού φτάσουμε σε αυτό, μια σειρά προβλημάτων πρέπει να επιληθούν πρέπει να δούμε ότι πρέπει να είναι ανταγωνιστικά τα ανανεώσιμα υπό οι ίσους όρους ε, και προϋποθέσεις όπως τα άλλα. Πρέπει να ενταχθούν στην αγορά. Πρέπει να πάψουν να υποστηρίζονται με επιδοτήσεις ε, και με δεκανίκια. Πρέπει μόνα τους αυθύπακτα αυτοτελώς να μπορέσουν να αναπτυχθούν. Διότι διαφορετικά αν δεν γίνει αυτό θα καταλήξουμε σε μια κατάσταση στην οποία οι δαπάνες που θα συνεπάγεται η υποστήριξη αυτή θα σημαίνει τεράστιες θυσίες και περικοπές. Για μας ε, το έλλειμμα το οποίο και υπερχρέωσης που έχει συσσωρευτεί όσον αφορά τις ε, ηλεκτρικές εταιρείες είναι 25 ή παραπάνω δις κιόλας ε, και αυτό είναι τεράστια ποσά. Λοιπόν, πρέπει να αρθούν τα εμπόδια ε, για την ε, προώθηση των ανανεώσιμων. Λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει κάθε δίκιο. Πρέπει να πάψουν να υπάρχουν επιδοτήσεις ε, για τα ορυκτά καύσιμα που ακόμα υφίστανται. Να μειωθούν οι γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις. Πρέπει να υπάρξουν ενιαίες θηρίδες. Πρέπει πολλά να γίνουν. Αλλά επίσης πρέπει να πετύχουμε μια ισορροπία μεταξύ της βούλησης να προωθούν τα ανανεώσιμα και της δυσκολίας να εξευρεθούν δημόσια κονδύλια και χρήματα για να γεφυροποιήσουμε το κενό που υπάρχει μεταξύ των παραδοσιακών πηγών ενέργειας και των ανανεώσιμων. Και επιπλέον για να είναι ανταγωνιστικά πρέπει να υπάρξουν κίνητρα για την τελειοποίησή τους και βελτιστοποίησή τους. Αφετέρου είναι αναγκαίο, απαραίτητο να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που συνεπάγονται τα ανανεώσιμα όσον αφορά την προσαρμογή των δικτύων. Όλοι γνωρίζουμε για τον χαρακτήρα τους αυτό που αυτό που είναι, ε, εποχη, είναι, είναι ε, εκ μια σειρά προβλημάτων πρέπει να αντιμετωπιστούν. Πολλές δράσεις ε, προαναγγέλλονται στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ιδιαίτερα η εμβάθυνση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς ενέργειας η συνεργασία στη Λεκάνη Μεσογείου, μηχανισμοί για τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών. Εκείνοι που έχουν πολλά ανανεώσιμα μπορούν να ε, αναζητήσουν συνεργασία με εκείνα που έχουν λιγότερο ανεπτυγμένα τα ανανεώσιμα. Ένα ευρύτατο φάσμα ενεργειών και δράσεων. Όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση για τα ανανεώσιμα και να συνεισφέρουμε. Αλλά πρέπει όλοι να συμφωνήσουμε ότι πολλά προβλήματα πρέπει ακόμα να επιληθούν για να τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ. Συνάδελφος Πίτερ παρακαλώ. Συνάδελφο, ή παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω ότι έχοντας ακούσει την παρέμβαση προηγούμενα των αξιότιμων ευρωβουλευτών που παρενέβησαν, για μένα δεν είναι αποδεκτό να επιδοτείται μόνο ένας τύπος, μια μορφή ενέργειας. Κατανοώ ότι δίνουμε και δώσαμε ειδικά κονδύλια και για την έρευνα ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης. Δεν μπορούμε να πούμε ότι μόνο οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πρέπει να αντλούν, μόνο τα ανανεώσιμα πρέπει να αντλούν κονδύλια και να μπορούν να υποστηριχθούν γιατί μπορεί να υπάρχουν και άλλες πηγές ενέργειας που να, βρεις, να έχουν μόνο εν μέρει ανακαλυφθεί και που δεν προάγονται ακόμα επαρκώς. Δεν μπορούμε μόνο να επικεντρωθούμε αποκλειστικά στα ανανεώσιμα και να αυταπατώμεθα. Οι τιμές αυτή τη στιγμή είναι απρόσθεσες για τους πολίτες μας και πρέπει κυρίως να, να δούμε τι θα γίνει με όλους τους πόρους, με όλες τις πηγές. Όχι μόνο τα ανανεώσιμα αλλά και με άλλες πηγές ενέργειας. Δεν μπορούμε έτσι ξαφνικά να πούμε ότι τα ορυκτά καύσιμα δεν θα μπορούν να εξεταστούν ως ε, δυνατότητα και να μην υπάρχει πλέον έρευνα. Πρέπει να υποστηρίξουμε την έρευνα και την καινοτομία. Δεν ξέρω, ίσως υπάρχει μια δυνατότητα, για να δώσω ένα παράδειγμα, με τα αέρια ε, σχιστολίθου, να χρησιμοποιήσουμε τις βέλτιστες ε, τεχνολογίες από πλευράς Ευρώπης για τα σχιστολιθικά αέρια, να μπορέσουμε να υποφεληθούμε από τα καλύτερα πλεονεκτήματα το παραδοσιακό, σε σχέση με το παραδοσιακό φυσικό αέριο. Δεν θα πρέπει να επικεντρωνόμαστε μόνο αποκλειστικά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δύο κράτη τα οποία δεν μπορούν να τα καταφέρουν με αυτή τη δυνατότητα. Πρέπει να δούμε τις γεωγραφικές μας δυνατότητες. Δεν μπορούμε όλοι παντού να εξαρτώμαστε και να βασιζόμαστε στην αιωλική ενέργεια δεν είναι δυνατό να υπάρχει μόνο μία πηγή ενέργειας για όλες τις χώρες αποκλειστικά. Δεν έχουμε δυνατότητα μετατροπής ή μετασχηματιστές, επαρκής μετασχηματιστές. Πρέπει σε διαφορετικές μορφές ενέργειας να θέσουμε το επίκεντρο, το κέντρο βάρους και όχι σε μία μόνο. Πρέπει να είμαστε ευφύης εναντί των πολιτών μας, να είμαστε αποτελεσματικοί και επαρκείς και αυτό πρέπει να δούμε πώς μπορεί να βελτιωθεί η ζωή των πολιτών μας μέσα από ο κύριος παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να σας πω ότι με εντυπωσίασαν αυτά που πρότεινε ο κύριος Τόμας, ε, δηλαδή ε, αυτό που είπε ότι οι τράπεζες της Κίνας δεν κερδοσκόπησαν. Δηλαδή εσείς τι κάνετε, πενεύετε την μετακομμουνιστική σκιώδη οικονομία, δηλαδή αυτό μας συστήνεται εδώ στην Ευρώπη, το φτηνό κεφάλαιο, περίεργα αυτά που λέτε, ενδιαφέροντα όμως. Κατά τα άλλα, το βρίσκω περίεργο το ότι η πράσινη πολιτική είναι εκείνη οι οποίοι παρεμποδίζουν τις λύσεις σε εθνικό επίπεδο. Οι πράσινοι είναι εκείνοι που εμποδίζουν την αγορά ε, των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια Και πραγματικά, ε, με πολύ μεγάλη αγωνία, περιμένω να δω τι θα κάνετε, πώ θα τα βρείτε με του συναντέλφου σα από τα άλλα εθνικά κοινοβούλια. Εγώ έρχομαι από μια περιοχή η οποία είναι αποτελεσματικότερη ε, στι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια από το Μούνστα. Εμεί δεν είμαστε ούτε παράκτη περιοχή, ούτε ορεινή, αλλά και από πλευρά το οποίο δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Είμαστε στο κέντρο τη Γερμανία. Αν πάτε στο Μούνστερλαντ θα δείτε ότι υπάρχουν παντού εκεί εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκές και υπάρχουν ε, και σπίτια ε, τα οποία απλά κατασκευάζονται για να υπάρχει στέγη για, τις, τα φωτοβολταϊκά. Αν πάτε στο Μίντερλαντ θα δείτε παντού δύο μάζα. Το 70% των καλλιεργιών είναι ε, καλαμπόκι. Κανείς πια δεν παράγει τρόφιμα. Στο βλέπετε ότι το 70% είναι ε, καλλιέργειες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για για την αιωλική ενέργεια. Και εμείς ε, στη Γερμανία ε, δυστυχώς ε, έχουμε αντιμετωπίσει με τεράστιο κόστος, ενώ από την άλλη υπάρχουν περιοχές που η ενέργεια μπορεί να είναι πολύ πιο φτηνή. Αυτή η ενέργεια είναι πάρα πολύ ακριβή που παράγεται σε εμά. Κανείς δεν μπορεί να την αγοράσει. Άρα δηλαδή η μόνη συνέπεια που προκύπτει, δυστυχώς δεν ακούσαμε εμείς την παρατήρηση Κοιτάξτε, ε, συμβατές ε, μορφές ενέργειας μόνο στο Λουξεμβούργο είναι περίτη η συμβατή ενέργεια. Παντού αλλού είναι απαραίτητη συμβατή ενέργεια, οι παραδοσιακές μορφές ενέργειας για να μπορεί κανείς να ανταπεξέλθει στη ζήτηση. Εγώ λοιπόν Είμαι πεπισμένο ότι χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή αγορά. Συνάδελφε Βιντάλ Κουάντρας, δεν χρειαζόμαστε μεγαλεπίβολα προγράμματα. Νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε και κάποια ευκαιρία στην αγορά να αυτοοργανωθεί. Γιατί αν ήταν δυνατόν να εισάγουμε φωτοβολταϊκή ενέργεια από την Νότια Ευρώπη, αν αυτό το επέτρεπε η γερμανική πολιτική, δηλαδή να εισάγεται βιομάζα από την Νότια Ευρώπη, αν ευρωπαϊκούς κανόνες για κάτι τέτοιο, αν ήταν δυνατό να προσφέρουμε ενέργεια μέσα από το κανάλι της Μάνχης, τότε ε, για μας η ε, διαρθρωτική πολιτική θα ήταν πολύ πιο φτηνή. Και επιτέλους ε, πρέπει να έχουμε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση, να γνωρίζουμε ότι η αγορά είναι καθοριστική σημασία για τις ανώσιμες πηγές ενέργειας, όχι η παροχή κεφαλαίου. Για αφήστε λιγάκι την αγορά να λειτουργήσει και θα δείτε πώς θα τα καταφέρει. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε κύριος ε, Μετσάρος έχει το λόγο. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε μόλις τώρα ο κύριος Πίπα. Πράγματι πρέπει επιτέλους ορμόμενοι από αυτήν την ε, εφορία η οποία προκύπτει από το ότι μιλάμε συνεχώς για τις ανώσιμες πηγές ενέργειας να προχωρήσουμε μπροστά. Ξέρουμε ότι οι ανανόσιμες πηγές είναι καθοριστική σημασία στο πλαίσιο του ενεργειακού μείγματος και κανείς δεν αμφισβητεί τη σημασία αυτών των πηγών ενέργειας. Όμως οφείλουμε να γνωρίζουμε αυτή δεν είναι η μοναδική λύση. Δεν πρέπει να αυτά πατώμεθα. Δεν υπάρχει μια πολιτική που να λύνει όλα μας τα προβλήματα. η ανταγωνιστικότητα είναι καθοριστική σημασία, η πρόσβαση στην ενέργεια, τεχνικές λύσεις που είναι απαραίτητες, ε, και οι δικές μας οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Αυτά είναι σημαντικά. Αν δούμε λοιπόν τις ανώσμες πηγές κάτω από αυτό το πρίσμα, ε, θα κατανοήσουμε ότι χρειαζόμαστε στα διάφορα κρατημέλη ένα ισορροπημένο ενεργειακό μείγμα. Ακούσαμε λοιπόν ένα παράδειγμα ότι όλες ε, οι κιλοβατόρες ενέργειας οδηγούν σε νέες θέσεις εργασίας. Κάθε κιλοβατόρα σε μία νέα θέση εργασίας. Καλό το επιχείρημα, αλλά οφείλουμε επίσης να κατανοήσουμε ότι αυτό δεν έχει μόνο ε, υπέρ, και κατά, διότι οδηγεί σε αύξηση του κόστους. Για μένα λοιπόν αυτό δεν είναι πιστικό επιχείρημα. Αν δούμε λιγάκι την κλιματική αλλαγή, διαπιστώνουμε ότι έχουμε μόνο δύο ε, πηγές ενέργειας ε, που μας στηρίζουν στον αγώνα μας, τη φωτοβολταϊκή και την αιωλική. Η βιομάζα απλά οδηγεί στο να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα όπως και στις ε, παραδοσιακές πηγές στα ορυκτά καύσιμα γιατί ε, σε τελική ανάλυση αυτό που κάνουμε είναι απλά να εκμεταλλευόμαστε τον άνθρακα που ε, βρίσκεται στο υπέδαφος εδώ και χιλιάδες χρόνια. Στην, ε, η βιομάζα δεν μας βοηθάει στο να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή και εκτός αυτού κάποιες αγροτικές εκτάσεις χρησιμοποιούνται για να παραχθεί βιομάζα, ούτε και αυτό βοηθάει. Άρα δηλαδή οφείλουμε να βρούμε νέες προσεγγίσεις. Χρειαζόμαστε όμως ένα ισορροπημένο ενεργειακό μείγμα. Η ενεργεια και οι ανανεώσιμες πηγές δεν αποτελούν πανάκια. Ε, εμπιστεύομαι ε, τον κύριο Ρόιλ. Ε, ξέρω ότι η έκθεση στα χέρια του είναι σε καλά χέρια. Ξέρω ότι θα συντάξει μια ισορροπημένη έκθεση. Και εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε για τη Γερμανία. Δηλαδή, αυτά που συμβαίνουν με τη Γερμανία, στη Γερμανία με την ολική ενέργεια οδήγησαν στο ότι επηρεάστηκε πάρα πολύ το ενεργειακό ηλεκτρικό δίκτυο στην Τσεχία. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε αυτά τα FEE δίκτυα, τα smart grids που αναφέρθηκαν. Και όσον αφορά τις ε, κρατικές επιδοτήσεις, οι διαφορές ανάμεσα στα διάφορα κρατημέλη είναι πολύ μεγάλες και δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε ένα κράτος μέλος να χορηγούνται επιδοτήσεις για κάποιες ενεργειακές μονάδες, ενώ σε άλλο κράτος μέλος να μην επιτρέπεται απολύτως τίποτα. Παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε δύο-τρία σχόλια. Είμαι πεπισμένος ότι το 2050, το 2100 πάντως σίγουρα, αλλά ίσως ήδη το 2050, οι πηγές ενέργειας στην Ευρώπη και στον κόσμο θα είναι όλες ανανεώσιμες. Ίσως υπάρχουν ακόμα κάποιες συμβατικές άνθρακας ή πυρηνική, αλλά είμαι πεισμένος ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και αυτό είναι ο μόνος δρόμος για το μέλλον. Δεύτερο, όταν αναλογίζεται κανείς τι ανανεώσιμες, μπορεί, μπορεί βέβαια να το κάνει κανείς στην κλίμακα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πρέπει να εξετάσει και σε κάθε περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ποια είναι η πρωταρχική πηγή ενέργειας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Εδώ είναι ο άνεμος, αλλού είναι η θάλασσα, αλλού είναι το βιολογικό αέριο ή ο ήλιος και ούτω καθεξής. Υπάρχουν πρωταρχικές ε, πηγές. Βέβαια, η εξι διαφορετικες πρωταρχικες πηγες είναι ο ήλιος, ακόμα και ο άνεμος είναι παράγωγο της ηλιοφάνειας. Αυτές λοιπόν τις ιδιαιτερότητες, τις περιφερειακές, πρέπει να εκμεταλλευτούμε για τις, ε, για τις ανανεώσιμες πηγές. Υποδομές. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητο να φτιαχτούν αυτοκινητόδρομοι ανανεώσιμων ενεργειών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μπορέσει να υπάρξει μια αναδιάρθρωση για το ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ πάντα βέβαια, για τη μεταφορά και τη διανομή του, αλλά στο τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο. Στο ευρωπαϊκό μου φαίνεται ότι αφενός είναι πολύ δαπανηρό, κάτι τέτοιο, αλλά και άχρηστο. Εν τέλει, επειδή δεν θέλω να μακρηγορήσω μια και τα είπε θαυμάσια ο κύριο Τουρμέ για τι επιχορηγήσει εδώ και μια πεντηκονταετία. α εξετάσουμε τα κεφάλαια που έχουν επενδυθεί στην ε, πυρηνική ενέργεια για να επιτύχουν τελικά απογοητευτικά αποτέλεσματα. Εγώ προτείνω λοιπόν τα επόμενα 50 χρόνια να επενδυθούν τα ίδια σε ποσά κεφάλαια στις ανανεώσιμες ενέργειες που θα αποδώσουν, πιστεύω, όχι απογοητευτικά αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Κράουσμαν. Κρότσμαν, συγγνώμη. Κύριε Τούρμε, στη Γερμανία ε, έχουμε το φαινόμενο, διακόπτει ο κύριος Τούρμες, δεν ακούμε όμως τι λέει, ότι έχουμε βραβεία για την ενέργεια, υπάρχουν και επιπτώσεις, όπως ξέρετε υπάρχουν προτάσεις οι αυξανόμενε τιμέ των ανανεώσιμων ενεργειών να μην επιβαρύνουν τα νοικοκυριά, διότι κάτι τέτοιο θα έχει δραματικέ επιπτώσει και στην Ευρώπη ω έδρα βιομηχανία. Γι' αυτό και πρέπει να σκεφτούμε. Δεν είναι κανεί εδώ αντίθετο με τι ανανεώσιμε ενέργειε, αλλά πώ μπορούμε να διαμορφώσουμε σωστά τη διαδικασία αυτή. Ακόμα δεν υπάρχει τρόπο αποδικευσή τη και γι' αυτό πρέπει να δούμε σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει ήλιος, δεν φυσάει ο άνεμος, να έχουμε και τότε ενέργεια, έτσι, για να μπορεί να συνεχίζεται η βιομηχανική παραγωγή. Και θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα το πετύχουμε αυτό. Δεν θέλουμε εμείς νέες επιχορηγήσεις. Γιατί είναι τόσο φτηνή η ηλιακή ενέργεια. Αφενός διότι επιχορηγείται, αλλά και β, δεύτερο, διότι στη Γερμανία εμείς έχουμε πολύ μικρές επιχειρήσεις. Είδα η Bosch να λέει ότι θέλει να μπει στην ηλιακή ενέργεια, αλλά χωρίς επιχορηγήσεις. Άρα χρειάζεται ισχυρές με, ε, ε, επιχειρήσεις με, με μεγάλα κεφάλαια, ισχυρές δηλαδή, που να μπορούν να μπουν στον ε, χώρο αυτό. Γι' αυτό χρειαζόμαστε, και αυτό υποστηρίζω τον κύριο Ρόιλ, μια ενεργειακή πολιτική ενδεχομένως και μια διασύνδεση, μια διαδικτύωση των διαφόρων προσφόρων που έχουμε. Και αν το επιτύχουμε αυτό, τότε θα έχουμε την ευκαιρία. Διότι δεν καταφέρουμε να έχουμε ενέργεια σε αποδεκτές τιμές, τότε η αποδοχή των νέων ανανεώσιμων ενεργειών θα μειωθεί σημαντικά. ...60% του κόστους για τη διοχέτευση ενέργειας από τα νοικοκυριά στα κεντρικά δίκτυα, 60% λοιπόν είναι διοικητικό κόστος. Αυτό λοιπόν δεν ενδιαφέρει του καταναλωτές, δεν είναι στο συμφέρον των καταναλωτών. Και όταν οι καταναλωτές δεν θα μπορούν πλέον να ανταποκριθούν στο κόστος, τότε θα πρέπει να, να μπει ε, μέσα και η βιομηχανία. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και δεν είναι σοβαρό όταν λέμε για 50% παραγωγή ενέργειας από την ε, ηλιακή ενέργεια. Εκεί όπου υπάρχει περισσότερος ήλιος, περισσότερος άνεμος, εκεί πρέπει να παραχθεί φθηνότερα και να έρθει μέχρι μας. Είναι και οι γραμμές, έχετε δίκιο βέβαια, πρέπει να υπάρξουν και οι γραμμές. Βέβαια, αποκέντρωση είναι ένα θέμα. Ε, εγώ είμαι υπέρ των μεγάλων αυτοκινητόδρομων τη ενέργειας, αλλά αποκεντρωμένα μόνο δεν επιλύεται το πρόβλημα και γι' αυτό χρειαζόμαστε του μεγάλου τους μεγάλους αυτοκινητόδρομους ενέργειας. Και γι' αυτό η πρόταση του Γερμανού Υπουργού ε, Ενέργειας με 5% δηλαδή από τα κέρδη της βιομηχανίας να πηγαίνουν στις επενδύσεις. Πολύ ωραία. Τελειώσαμε λοιπόν την ε, όλη συζήτηση και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ και καλησπέρα σας. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προσβλέπει στην έκθεση αυτή. Ήδη ετέθησαν πολλά και σημαντικά θέματα. Φερθεί και στην έκθεση Επιτροπής. Όπως και εσείς στην έκθεση αναφέρουμε γιατί πρέπει να προαχθεί η να προαχθούν οι ανώσιμες πηγές για να αντιμετωπιστούν οι διακυμάνσεις στις τιμές των ορυκτών καυσίμων ή για να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι ή αν θέλετε και για να δοθούν κίνητρα στην ανάπτυξη, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η ανακοίνωση της Επιτροπής επισημαίνει το στοιχείο του κόστους και επίσης αναφέρει ότι υπάρχουν πάρα πολλά που μπορούμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε το κόστος. Όσο λοιπόν πιο δύσκολη είναι η οικονομική κατάσταση, τόσο πιο σημαντικό είναι να ε, επιδιώξει κανείς την επίτευξη των στόχων και να προάγει τις ανανόσιμες πηγές. Γι' αυτό λοιπόν εμείς θέλουμε να εκπονήσουμε κατευθυντήριε γραμμές για το πώς μπορεί να υπάρξει η σύγκληση ανάμεσα διάφορα κρατημέλη. Όχι απαραίτητα εναρμόνιση, γιατί πρέπει να παραμείνει ένα σταθερό περιβάλλον επενδύσεων, αλλά υπάρχει περιθώριο έτσι ώστε τα κρατημέλη να μάθουν το ένα από το άλλο, να εισάγουν βέλτιστες πρακτικέ, ε, μηχανισμού ε, για να εμφανιστούν οι ενώσιμες πηγές στην αγορά και όλα αυτά τα μέτρα έχουν ήδη παρουσιαστεί από τα κράτη-μέλη. Ήδη υπάρχουν, ε, υπάρχει κάποια μετακίνηση από το feed-in tariffs στο feed-in premiums. Ε, θεωρούμε ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης ε, τα μέτρα στήριξης ε, μπορούν να είναι αποτελεσματικά. Η νέα οδηγία έχει ε, βοηθήσει στο να δημιουργηθούν οι μηχανισμοί εκείνοι έτσι ώστε οι ενώσιμες πηγές να είναι αποτελεσματικές στη σχέση κόστος-οφέλους παντού, όχι μόνο στα κράτη-μέλη. Η Κομισιόν επίσης προτίθεται να εκπονήσει κατευθυντήριες γραμμές στους μηχανισμούς συνεργασίας έτσι ώστε να βελτιωθεί ε, η σχέση κόστους-οφέλους πάντα σε σχέση με τις ανανεώσιμες πηγές στην Ευρώπη. Αναφερθήκατε και σε ανάγκες ε, υποδομής. Υπάρχει το σχετικό πακέτο που αυτή τη στιγμή πρόκειται να εγκριθεί, καλό να εγκριθεί γρήγορα για το μέλλον των ανανόσιμων πηγών, αλλά πρέπει να έχουμε κατά νου και τα δίκτυα διανομής και τα ευφύ δίκτυα, γιατί και αυτά θα παίξουν ρόλο στο να διευκολύνουν την, το, την ε, των ανανεώσιμων ε, στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Υπάρχει λοιπόν, υπάρχουν όλα αυτά, η υποδομή, η εσωτερική αγορά. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι οι αλλαγές που θα κάνουμε θα βοηθήσουν τον ενεργειακό τομέα. Υπάρχουν πολλές δυνάμεις που έχουν ως στόχο να επιβραδύνουν την αλλαγή στον τομέα αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς ε, πλέον ε, μετακινούμεθα ε, λόγω της κλιματικής αλλαγής και γι' αυτό πρέπει να διασφαλίσουμε οι αλλαγές που κάνουμε πράγματι προάγουν την αλλαγή και δεν μας πάνε πίσω στον 20ο αιώνα. Η όλη ιδέα είναι ότι ε, θα πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα προς το μέλλον, προς αυτές τις ιδέες, έτσι ώστε ε, να ε, συνεχίσουμε να εκμεταλλευόμαστε την ενέργεια με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργούνται θέσει απασχόλησης. Να επιτευχθούν οι στόχοι μας και αυτό να γίνεται με έναν τρόπο αποτελεσματικό, πάντα από το πρίσμα της σχεση κοστους κόστους-οφέλους. Ο κύριος Ρόιλ τώρα έχει το λόγο για να ανακεφαλαιώσει. Κύριε Ρόιλ, πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα είμαι πολύ σύντομο τώρα ολοκληρώνοντα και τελειώνοντα για απόψε. Πρώτον, θέλω να παρακαλέσω τα θέματα στα οποία έχουμε κάποιε τριβέ ή ε, είναι αμφίσιμα να τα βάλουμε σε παρένθεση, να τα αφήσουμε εκτό. Αν και πόσο, ποια είναι η σημασία των άλλων πηγών ενέργεια. Α προσπαθήσουμε να τα αφήσουμε στο περιθώριο Ποιος φταίει για το ότι βρισκόμαστε τώρα σε μια τέτοια κατάσταση. Εκεί τώρα, αυτά σε παρένθεση. Και να δούμε πώς μπορούμε να τα καταφέρουμε από κοινού. Να πούμε, η κατάσταση είναι δεδομένη και έχει ως έχει. Συμφωνούμε ότι οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια πρέπει να έχουν ένα, μέσο, ένα μέλλον, μεγάλε, μικρέ και τα λοιπά, άσχετα. Με ποια μέσα μπορούμε να καταφέρουμε να πετύχουμε τις βέλτιστες επιπτώσει, να κρατήσουμε τι δαπάνε χαμηλά, σε χαμηλά επίπεδα και να είμαστε αποδοτικοί και να έχουμε τι καλύτερε επιδόσει. Αυτά να κάνουμε. Όλα τα άλλα τα βάλουμε σε μια παρένθεση, στο περιθώριο να μην έχουμε αντιπαραθέσει, σε αυτά να επικεντρωθούμε και να προσπαθήσουμε να τα πετύχουμε και να τα καταφέρουμε σωστά. Δεν μπορεί κανεί μέσα σε ένα πλαίσιο σαν αυτό να τα καταφέρει όλα τα επιπαντό του επιστητού να τα επιλύσει. Η αρμοδιότητα και περισσότερε εξουσίε που χρειαζόμαστε ευρωπαϊκά. Εν πάση περιπτώσει, αν συμφωνήσουμε επ' αυτόν, μπορούμε να δούμε σε αντιπαράθεση σε, ε, έναντι του Συμβουλίου τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτή είναι η προσπάθεια, το εγχείρημα. σω τα καταφέρουμε από κοινού όλοι ενωμένοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Ρόιλ. Θα ήθελα να σας πω ότι προβλέπεται και ένα σχετικό εργαστήριο στις 18 Νοεμβρίου από τις 15 έως τις 18 ε, και εκεί θα συζητηθεί αυτή η έκθεση. Επίσης ε, και θα συζητηθεί και στις 28 και στις 29 Νοεμβρίου. Σας ευχαριστώ. Πάμε τώρα στο επόμενο σημείο της μερίσιας διάταξης που αφορά την παρουσίαση από την Επιτροπή των εκτελεστικών πράξεων για τον κανονισμό του roaming. Για να δούμε πού ακριβώς βρισκόμαστε. Η Επιτροπή έχει το λόγο, ο κύριος Τεράβα, για να μας παρουσιάσει την κατάσταση. Thank you, Madam Chair. Uh, yes, indeed, uh, my intention is to give you... Ευχαριστώ. Θα σας ενημερώσω για το που βρίσκεται η Κομισιόν με την ε, εφαρμοστική πράξη για τις υπηρεσίες περιαγωγής. Όπως θα θυμάστε, ο κανονισμός περιαγωγής που εγκρίθηκε τον Ιούνιο περιλαμβάνει χωριστές υπηρεσίες πώλησης ε, υπηρεσιών περιαγωγής. Προβλέπει δύο υποχρώσεις αφενός τους εγχώριους παρόχους να δίνουν τη δυνατότητα στους ε, πελάτες τους να έχουν πρόσβαση στις, σε μια δέσμη υπηρεσιών περιαγωγής, SMS κλπ. Και δεύτερο, ο κανονισμός επιβάλλει την υποχρέωση παρόχων υπηρεσιών εγχωρίων και περιαγωγής να μην εμποδίζουν τους πελάτες τους να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες περιαγωγής που προσφέρει άμεσα ένα δίκτυο υποδοχής, σε άλλη χώρα δηλαδή. Ο, στο άρθρο 5 ο κανονισμός απαιτεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγκρίνει πράξεις εφαρμογής που να περιέχουν τις λεπτομέρειες για την ξεχωριστή πώληση καθώς και πληροφορίες για τις σχετικές ενημερώσεις, τις απαιτήσεις ενημέρωσης δηλαδή, που θα πρέπει να δίνουν οι πάροχοι, οι εγχώροι πάροχοι στους περιαγόμενους ε, πελάτες. Στη βάση αυτή, το καλοκαίρι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέτασε τις διάφορες τεχνικές λύσεις για την εφαρμογή αυτής της χωριστής πώλησης, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραλλαγές, τις οποίες γνωρίζουν όσοι συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή, όταν συζητήσαμε δηλαδή τον κανονισμό περιαγωγής. Μιλήσαμε τότε για λύσεις όπου λέγονται Dual EMC και Single EMC και LBO. Αυτά είναι τα αρχικά στα αγγλικά. Αφού λοιπόν συζητήθηκαν οι τεχνικές αυτές λύσεις σε αντιπαραβολή με τα κριτήρια του άρθρου 5 του κανονισμού περιαγωγής όπως ευχρηστία από πλευράς κατανολωτών, ε, χαμηλό κόστος καθώς και άλλα κριτήρια τα οποία έπρεπε να ικανοποιούν όλες οι τεχνικές λύσεις. Όμως τα κριτήρια αυτά σημαίνουν, και αυτό ήταν και το συμπέρασμα μεταξύ άλλων, ότι δεν υπάρχει μία και μοναδική τεχνική λύση η οποία να πληρεί όλα τα κριτήρια. Για το λόγο αυτό καταλήξαμε σε μία λύση που συνδυάζει και αυτό προβλέπεται στο άρθρο 4 προβλέπει συνδυασμό λύσεων που επιτρέπουν στον περιεχόμενο πελάτη να έχει πρόσβαση στις ε, υπηρεσίες περιαγωγής αλλά και εγχωρίως και στις χώρες, στις αγορές δηλαδή υποδοχής. Με μια βασική μορφή η λύση αυτή αποτελεί μια λύση αναπόλυσης, resale, που αυτό θα είναι σημαντικό για να διακριθεί και η κυριότητα της υπηρεσία από το δίκτυο. και επίσης η τεχνική λύση που επιτρέπει στους πελάτες να έχουν πρόσβαση ευθέως στις υπηρεσίες περιαγωγής του δικτύου της χώρας υποδοχής, χώρας όπου μεταβαίνουν δηλαδή και το λεγόμενο Local Breakout, LBO, που θα είναι η άλλη λύση. Έτσι λοιπόν προτείνουμε ε, συνδυασμό της Single EMC και της Basic LBO δύο αυτές τις τεχνικές λύσεις. Σύμφωνα με τον κανονισμό περιαγωγής έπρεπε να ζητήσουμε τη γνώμη του Οργανισμού των Ευρωπαίων Ρυθμιστών για το σχέδιο. Το πράξαμε τον Αύγουστο και την προηγούμενη εβδομάδα ο οργανισμός αυτός που λέγεται BEREC υπέβαλε τη γνωμοδότησή του για το Separate Sale και κατέληξε ότι ο συνδυασμός του Single EMC και του Basic LBO είναι η καλύτερη στην πραγματικότητα τεχνική λύση τουλάχιστον επί της παρούσης. Ο οργανισμός Μπέρεκ τόνισε επίσης ότι συνεχίζεται η τεχνολογική εξέλιξη και η εξέλιξη της αγοράς και ότι αυτό πρέπει να συνεχίσουμε να το παρακολουθούμε την εξέλιξη αυτή και αν αυτό καταστεί απαραίτητο να επανεξετάσουμε τις τεχνικές αυτές λύσεις αν όντως δηλαδή είναι και μακροπρόθεσμα οι προτιμότερες. Για το λόγο αυτό στο σχέδιο του εφαρμοστικού κανονισμού προβλέπουμε ότι όταν θα γίνει η επανεξέταση του κανονισμού περιαγωγής το 2016, ταυτόχρονα θα αξιολογήσουμε εάν όντως η τεχνική λύση που προτείνουμε χρειάζεται ίσως να προσαρμοστεί εν ώψη των εξελίξεων στην αγορά αλλά και στην τεχνολογία. Το κύριο σημείο εδώ είναι ότι με τον εφαρμοστικό κανονισμό πρέπει να δώσουμε σαφήνεια στον κλάδο για το τι πρέπει να εφαρμοστεί έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ε, συνεπή, συνεκτική και ταυτόχρονη εφαρμογή και στις 27 χώρες μέλη. Αυτό είναι μια πρώτη και σημαντική πτυχή του εφαρμοστικού κανονισμού. Τώρα, εάν αυτός ο κανονισμός, όπως τον προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εγκριθεί εν τέλει, είναι σαφές ότι οι λύσεις που ανέφερα προηγουμένως, Single EMC και Basic LBO, είναι αυτές που θα εφαρμοστούν. Υπάρχει και το θέμα βέβαια, που ίσως είναι και πιο σημαντικό, πώς δηλαδή θα πρέπει να εφαρμοστούν οι τεχνικές αυτές λύσεις. Εδώ υπάρχει ένας αριθμός τεχνικών απαιτήσεων από τα interface και θέματα τυποποίησης και ούτω καθεξής. Εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν επιθυμεί να επισέλθει ιδιαίτερα στις τεχνικές λεπτομέρειες στον εφαρμοστικό κανονισμό που είναι κάπως άκαμπτο κείμενο. Γι' αυτό θα περιοριστούμε μονάχα στην καταγραφή των βασικών απαιτήσεων που πρέπει να καλύπτουν οι τεχνικές λύσεις. Ταυτόχρονα, όπως είπε και ο οργανισμός Μπέρεξ στην ομοδότησή του, θα συνεχίσει να εκπονεί παραπέρα guidelines που θα περιλάβουν περισσότερες λεπτομέρειες για τις τεχνικές λύσεις. Ταυτόχρονα υπάρχει και μια απέτηση προς τον κλάδο, τον ίδιο, να συμφωνήσει επί ορισμένων πραγμάτων. Για παράδειγμα, τεχνικά interface. Πολύ τεχνικά θέματα αυτά, τόσο τεχνικά που είναι καλύτερο να συμφωνήσει επάνω σε αυτά ο ίδιος ο κλάδος, δηλαδή τα μέλη του κλάδου μεταξύ, του, τους. Ο κανονισμός προβλέπει υποχρέωση των παρόχων περιαγωγής να συμφωνήσουν επί των τεχνικών αυτών λεπτομεριών για τα interface ταυτόχρονα, ζητεί από τον κλάδο να συνέλθει και να ε, εγκρίνει μία πλατφόρμα όπου θα συζητηθούν οι λεπτομέρειες αυτές και όπου θα ε, παρακολουθούν οι συζητήσεις αυτές και η Κομισιόν και ο Μπέρεκ. Ένα σημαντικό στοιχείο είναι ο χρόνος. Όπως θα θυμάστε, η χωριστή πώληση υποτίθεται θα αρχίσει να εφαρμόζεται και θα είναι στη διάθεση των πελατών περιαγωγή από τον 7ο του 2014. Άρα δεν υπάρχει πολύ χρόνος μέχρι ότου ο κλάδο να υποχρεούται να θέσει σε εφαρμογή τα συστήματα και έτσι να ανταποκριθεί στην ημερομηνία στόχο. Έτσι πριν ήδη εγκριθεί ο εφαρμοστικός κανονισμός υπάρχει ανάγκη και ο Μπέρεκ από τη μια μεριά αλλά και ο κλάδος βεβαίως υπό το φως των συζητήσεων για τον εφαρμοστικό κανονισμό και για τις guidelines του Μπέρεκ να συνεργαστούν ώστε να προκύψουν και να μπορούν να εφαρμοστούν οι απαραίτητε τεχνικέ λύσεις ήδη από την 1η Εβδόμου 2014. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την παρουσίαση της ε, κατάστασης. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Νίμπλα που είναι η συγγητριά μας για την περιαγωγή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω θερμά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όλα αυτά που μας είπε και το βρίσκω πολύ καλό γεγονό ότι βρίσκεται σήμερα εδώ και παρουσιάζει μια ενδιάμεση έκθεση για το στάδιο εφαρμογής του κανονισμού περί δεν έχω και πολλές ερωτήσεις, διότι νομίζω ότι η διαδικασία τρέχει ακόμα. Η σύσταση Μπέρεκ ε, υπάρχει, η Κομισιόν έχει τοποθετηθεί επ' και ως ε, Κοινοβούλιο πρέπει να πούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τις δικές μας τις ε, πολιτικές επιταγές. Αυτό ε, δεν είναι κάτι ε, που θα το αποφασίσει το Κοινοβούλιο. Η ουσία βρίσκεται στη ΣΥΣΑ Συμπέρεκ και στην Κομισιόν. Πάντως χαίρομαι πάρα πολύ που μας ενημερώσατε για τις τεχνικές δυνατότητες. Και έχω το εξής ερώτημα. Θεωρείτε ότι το 2014 στην καταληκτική αυτή ημερομηνία θα έχουν οι πολίτες ε, τη δυνατότητα να αγοράζουν τα, ε, τις υπηρεσίες ε, περιαγωγής ξεχωριστά από τον δικό τους τον πάροχο. Δεν ξέρω, από ό,τι γνωρίζω εσείς έχετε κάποιες συζητήσεις με τους αρμόδιους βιομηχανικούς κύκλους. Πάντως ως επιλογή αυτό θα μπορεί να προσφέρεται το 2014. Και έχω και άλλη μια ερώτηση που δεν έχει σχέση με την εφαρμογή, αλλά είναι σημαντική για μένα. Μετά την 1η Ιουλίου του 2012, εγώ πήρα κάποια mail από κάποιους πολίτες που λένε, διάβασα στην εφημερίδα ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή ε, η περιεγωγή 17 cent ανά μεγαμπάιτ, αλλά εγώ δεν είδα να ισχύει αυτό στο δικό μου τον πάροχο. Ε, μάλιστα, το αντίθετο, ε, εντάξει, μειώθηκαν οι τιμές, αλλά ερωτώ εσάς Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μήπως εσείς πήρατε κάποιες διαμαρτυρίες ή ξέρετε καθόλου ε, τελικά ε, αν οι πάροχοι τήρησαν αυτά τα, αυτά τα νέα τιμολόγια ή μήπως υπήρξαν και σε εσά διαμαρτυρίες ε, ότι οι πάροχοι δεν εφαρμόζουν τις νέες, τα νέα τέλη όπως προβλέπεται στην οδηγία περί περιαγωγής που αποφασίστηκε από τον Ιούλιο. Κοιτάξτε, και μένα το ίδιο με απασχολεί συμφωνώ με αυτά που είπες και ε, θέλω και εγώ να ρωτήσω ακριβώς το ίδιο την Επιτροπή. Ε, ο λόγος ε, στην συνάδελφο. Προ λίγων εβδομάδων εγώ οργάνωσα με τον κύριο Τσίζεστερ μια ημερίδα ενημέρωσης όπου τέθηκε το θέμα αυτό και τον... Ε, της κινητής τηλεφωνίας δηλαδή και για την Ολλανδία όπου ο κυριότερος πάροχος για κάποιο άγνωστο λόγο έχασε ε, την πρόσβαση για κάποιο διάστημα και τώρα λέμε ότι υπό εξαιρετικές περιστάσεις θα πρέπει να μοιράζονται το δικτυό τους όταν δηλαδή εκπίπτει ένα μεγάλο μέρος του δικτύου να μοιράζονται οι διάφοροι πάροχοι ώστε να είναι πιο ε, ενισχυμένο το δίκτυο ή να υπάρχει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα του δικτύου. Αυτό μπορεί να γίνει ή υπάρχουν δυσκολίες αναλόγως με τη χώρα. Γιατί βρίσκω ότι η ανθεκτικότητα του δικτύου είναι σημαντική και για τους τελικούς καταναλωτέ, αλλά βέβαια και για τις επιχειρήσεις οι οποίες χρησιμοποιούν τα δίκτυα της κινητής τηλεφωνίας. Ε, δεν ξέρω αν θέλει και κάποιος άλλος να ζητήσει το λόγο. Αν ε, δεν υπάρχουν, ε, θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ε, απαντήσει στις ερωτήσεις που έθεσε η κυρία Νίμπλερ και όλοι οι άλλοι. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, καταρχήν εμείς ανέκαθεν πιστεύαμε αυτό που κάνουμε. Δηλαδή, ανέκαθεν πιστεύαμε ότι οι τεχνικές λύσεις είναι θα μπορούν να εφαρμοστούν μέχρι τα μέσα του 2014. Όπως σας είπα, είναι πολύ σημαντικό να υπάρξουν κάποιες εξελίξεις και γι' αυτό ε, όπως επίσης ε, και σχετικά με τον Μπέρεκ, οι ε, βιομηχανικοί κύκλοι εξετάζουν τις λεπτομέρειες, το πώς μπορούν να εφαρμοστούν αυτές οι λύσεις. Γι' αυτό λοιπόν για τον, τον Μπέρεκ και την βιομηχανική πλατφόρμα όλοι οι μετέχοντες ε, παίζουν σημαντικό ρόλο. Επίσης ε, δεν υπάρχει πολύς χρόνος. Αυτός ε, είναι ένας από τους λόγους γιατί χρησιμοποιήθηκε ως τεχνική λύση και το single MC γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να εφαρμοστεί από το dual MC. Είμαστε λοιπόν πεπισμένοι ότι όλα αυτά θα λειτουργήσουν θαυμάσια, αλλά βεβαίω για να γίνουν όλα αυτά είναι σαφέ ότι θα πρέπει να δεσμευτούν όλοι άμεσα ενδιαφερόμενοι. Τώρα, όσον αφορά την εφαρμογή των νέων κανόνων, οφείλω να ομολογήσω ότι δεν έχω δει να υπάρχουν πολλά παράπονα. Πήραμε κάποια παράπονα Αυτά ε, τα παραπέμψαμε στην Εθνική Ρυθμιστική Αρχή για να ελέγξει την κατάσταση, αφού αυτό είναι ο ρόλος της, αλλά σε σχέση με το παρελθόν ε, η περιαγωγή υπάρχει αρκετό καιρό και έχουν περιστεί οι διαμαρτυρίες. Και δεν μπορώ να πω ότι οι νέοι κανόνες προκάλεσαν ε, νέο ρημαγδό καταγγελιών. Πάντως, αυτό είναι κάτι που το Μπέρεκ παρακολουθεί και έτσι όταν ε, θα δημοσιευτεί η επόμενη έκθεση συμβατότητας θα δείτε ακριβώς ποια είναι η κατάσταση. Πάντως ε, η αλήθεια είναι ότι εμείς ε, επαγρυπνούμε και πρέπει να επαγρυπνούν βεβαίως και οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές για να διασφαλίζουν τη συμβατότητα. Τώρα, Όσον αφορά το θέμα της αντεκτικότητας, ε, το περιβάλλον θα πρέπει να διασφαλίζει την ε, προστασία των προσωπικών δεδομένων, την ασφάλεια και την ακαιρεότητα των ε, δικτύων, ότι αυτά γίνονται σεβαστά. Αυτά έμεσα ελήφθησαν υπόψη όταν επιλέξαμε την βέλτιστη τεχνική λύση. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς, ε, το λόγο λοιπόν, ε, κυρία Νίμπλερ, για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση, θέλετε να παρέμβετε. Κυρία Νίμπλερ, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Δεν έχω πολλά πράγματα να προσθέσω. Ευχαριστώ και πάλι για τις πληροφορίες. Και ελπίζω απλά ότι τώρα γοργά η υλοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα ακολουθήσει ώστε οι πολίτες μας στις χώρες μας να υποφεληθούν από αυτή την προσφορά της υπηρεσίας περιαγωγής από τον Ιούλιο 2014 να μπορέσουν να, να τις χρησιμοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο. Ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να τα εφαρμόσουμε όλα αυτά όπως πρέπει. Από τα όσα ακούσαμε δείχνουν όλα ότι πορεύονται προς τη σωστή κατεύθυνση. Και αν και μέχρι τα τέλη του έτους έτσι προχωρήσουμε, αυτό θα είναι κάτι το οποίο θα είναι καλό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε έτσι λοιπόν. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξή μας αφορά την ε, διάσκεψη, παγκόσμια διάσκεψη του Δεκεμβρίου για τις διεθνείς τηλεπικοινωνίες. Δεν, μπορεί σήμερα να, ε, το, δεν μπορούμε να το δούμε σήμερα γιατί από πλευρά αρμοδίων δεν, δεν παρίστανται. Έχουμε ξεπεράσει το χρόνο μας. Θα ήθελα για τα διάφορα να πω κάτι τώρα και σε σχέση με αυτό να πω ότι οι συμβαλόμενοι για την ε, για τις κλιματικές αλλαγές θα πρέπει σήμερα να ενημερωθεί αυτό το θέμα, να υπάρξει ενημέρωση με την κυρία Ούσκογκ ως εισηγήτρια, μπορούμε να το κάνουμε λοιπόν. Γνωρίζετε σχετικά ότι από πλευρά εισηγητού και σκιώδους εισηγητού και από πλευρά των μελών της κοινοβουλευτική Επιτροπής θέλουμε να συνεισφέρουμε ως Κοινοβουλευτική Επιτροπή με τα όσα προετοιμάσαμε για το ψήφισμα Ήτρε και Ένβη από πλευρά Ευρωκοινοβουλίου. Και αυτό το θέμα την προπαρασκευή δηλαδή για, το, για την ΚΟΠ έχει δοθεί εντολή και αποκινούμε την Επιτροπή Περιβάλλοντος να διαδραματίσουμε ένα ρόλο. Και έχουμε και τροπολογίες, κυρία Σαρτόρη, η πρόεδρός μας, όλα αυτά με μια επιστολή τα ανέφερε στον πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος, επιστολή που απεστάλλει. Έχετε λάβει αντί, αντίτυπα των τροπολογιών, έχετε ενημερωθεί. Θέλουμε να δούμε αν υπάρχουν αντιρρήσει ή όχι, αν μπορούμε να εγκρίνουμε λοιπόν τα σχετικά. Θα ήθελα επ' αυτού να δώσω τον λόγο σε κάποιο συνάδελφο. Ποιος θα είναι αυτός? Μάλιστα. Δεν μπορέσατε να ε, παρακολουθήσατε δεν προσέχατε. Κυρία Ούσκογκ, θα μπορούσατε να επεξηγήσετε αυτή την επιστολή, αυτή που αφορά και τις τροπολογίες μας και που προετοιμάστηκε με τις τροπολογίες και με τους κοιόδης εισηγητές της Κοινοβουλευτικής μας Επιτροπής, ώστε η Επιτροπή Ήτρε να συμμετάσχει στην προπαρασκευή του, της πρότασης ψηφίσματος και να έχει και εκείνη την επιρροή που θα μπορέσει να ασκήσει. Θέλετε να πείτε δύο λόγια γι' αυτό και για τις ε, τροπολογίες. Έχετε τον λόγο παρακαλώ. Ε, ε Σας ευχαριστώ πολύ Πατρίσια. Και εγώ προσωπικά θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στους σκιώδεις εισηγητές που ενεπλάξαν και συμμετείχαν σε αυτό το έργο. Και όπως και συνέβη και σε προηγούμενα άλλα χρόνια, είχαμε στεναρή βούληση και από πλευρά της Επιτροπής Βιομηχανίας και της Επιτροπής Φυσικά Περιβάλλοντος, ώστε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία, ώστε με βάση αυτή να μπορέσουμε να έχουμε κοινέ θέσεις με τις οποίες θα καταλήγαμε στην διάσκεψη για το περιβάλλον, για τα περιβαλλοντικά θέματα και τις κλιματικές αλλαγές. Είναι γνωστό ότι υπάρχει δυσκολία να επιτευχθεί από τη συμφωνία δεδομένων όλων αυτών των θεμάτων και ως κοινοβούλιο θα πρέπει κάπου να καταλήξουμε προσερχόμενοι σε αυτή τη σύνοδο. Πέρυσι γνωρίζετε ότι διεξήχθη στο Ντέρμπαν αυτή η συζήτηση της Νότιας Αφρικής και διαδραμάτισε η Ένωση ένα μεγαλύτερο, πιο σημαντικό ρόλο σε σχέση με το παρελθόν. Πολλές από τις άλλες χώρες που συμμετείχαν έστρεψαν το βλέμμα και πρόσεξαν ιδιαίτερα να κατανοήσουν ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι λοιπόν ήρθε η χρονική στιγμή να επαναλάβουμε αυτό το εγχείρημα. Έχουμε συνδυάσει μια χειροπιαστή, πραγματιστική, ρεαλιστική προσέγγιση με τους στόχους για τις κλιματικές αλλαγές επί των οποίων είχαμε επιτύχει συμφωνία. Δύο βαθμοί ε, μέγιστη αύξηση της ε, θερμοκρασίας του περιβάλλοντος. Ε, θέλουμε να συνδυάσουμε όλες αυτές τις προσπάθειες σε σχέση με τους στόχους που συμφωνήθηκαν σε επενδύσεις σε, αηφόρα, σε ένα αηφόρο χρονοορίζοντα των δράσεών μας για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών αλλαγών. Αυτά είναι τα πράγματα στα οποία συμφωνήσαμε σε σχέση με το έγγραφο που μπορείτε να διαβάσετε. Ε, σας ευχαριστούμε και εμείς ε, και βεβαίως ε, επειδή δεν υπάρχουν αντιρρήσεις γκρίνεται αυτή η επιστολή που στάλε από τον κύριο Σαρτόρη. Νομίζω ότι ήρθε η κυρία Ρίτσορτς. Τώρα δεν ξέρω να δώσω εγώ τις πληροφορίες. Λοιπόν, να σας ενημερώσω όσον αφορά τις αποφάσεις που λήφθησαν σήμερα το πρωί στις συνεδρίες των συντονιστών. Και οι αποφάσει που λήφθησαν είναι οι εξή. Ε, θα υπάρξουν αντιπροσωπείε τη Επιτροπή ε, Ήτρα το 2013 στην ε, Νότιο Κορέα, στην Ιαπωνία και ένα Internet Governance Forum το οποίο θα λάβει χώρα στον Μπακού. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πάμε στη Λουθουανία, στην Ελλάδα στην ε, Σεβίλη. Αυτή θα είναι η τρίτη αντιπροσωπεία που θα πάει εκεί. Θα υπάρξουν ε, πέντε ακροάσεις ε, για πάρα πολλά θέματα, τα οποία θα σας παρουσιαστούν λεπτομερώς γραπτά, κατόπιν ε, θα θυμάστε για τις δημόσιες ακροάσεις. Μία θα λάβει ακόμα χώρα το 2012, αφορά στην ε, προστασία των ε, δεδομένων στις 17 Δεκεμβρίου και η άλλη το clouding computing Ιανουάριο-Φεβρουάριο του επόμενου έτους αλλά θα πρέπει να ξεκινήσουμε ήδη αμέσως τώρα τις προετοιμασίες τη σιδηρουργία. για τη σιδηρουργία θα υπάρξει προφορική ερώτηση ε, η οποία θα κατατεθεί τον Νοέμβριο σε αυτή την Ολομέλεια. Και όσον αφορά ε, τις εκθέσεις για το cloud computing στην Ευρώπη, η έκθεση θα γίνει από το ΕΛΚ, θα υπάρξει κατόπιν μία γνωμοδότηση ε, για την Ευρώπη και θα υπάρξει και ένα σχέδιο πρότασης το για τα πυρηνικά, το οποίο επίσης ε, και γι' αυτό θα υπάρξει προφορική ερώτηση. Αυτές είναι οι βασικές αποφάσεις που ελήφθησαν ε, σήμερα το πρωί. Και νομίζω ότι μπορούμε να ε, ρωτήσουμε το λέω αυτό για να μεταφραστεί, να απευθυνθούμε στη γραμματεία και να ζητήσουμε οι εκπρόσωποι της Επιτροπής που έρχονται εδώ να έχουν την καλοσύνη να φτάνουν ένα τέταρτο νωρίτερα ε, γιατί με τον τρόπο αυτό ε, μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη ευελιξία. Δεν χρειάζεται δηλαδή να φτάνουν στο παραπέντε, να φτάνουν λίγο νωρίτερα παρακαλώ. Και νομίζω ότι μπορούμε να διακόψουμε για λιγάκι ε, αν δεν υπάρχει καμιά αντίρρηση. Επόμενη συνεδρίαση στις 5 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες. Qualche minuto di attesa, se να δούμε αν έρχεται η κυρία Ρίτσο. qualche minuto nell'attesa che appunto facciamo un ultimo coup de fil a Madame Richards. Θα περιμένουμε λίγο να δούμε αν έρθει η κυρία Richards. Φτάνει, φτάνει μας.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 Eh, Μου λένε ότι δεν έχει φτάσει ακόμα η κυρία Ρίτσαρτς. Εγώ λοιπόν προτείνω το εξής. Αν ε, συμφωνείτε κι εσείς. Η ενημέρωση που πρέπει να μας κάνει η κυρία Ρίτσαρτς για την προετοιμασία της παγκόσμιας διάσκεψης για τις τηλεπικοινωνίες που θα λάβει η χώρα το 2012 που στη Τόρχα Α, στο Ντουμπάι. Στο Ντουμπάι αυτή η ενημέρωση θα είναι αντικείμενο μιας γραπτής ενημέρωσης που θα σταλεί σε όλα τα μέλη της Επιτροπής και έτσι θα μπορούμε και εμείς να κάνουμε τις παρατηρήσεις μας. Όπως σας είπα, ε, πρόκειται για την ε, προετοιμασία σε αυτή την ε, σημαντική διάσκεψη. Έτσι λοιπόν θα έχουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να μπορέσουμε και εμείς να ε, προσθέσουμε την δική μας την άποψη. Όπως σας είπα θα τα πούμε στις 5 Νοεμβρίου. Κλείνουμε τελείωσαν οι εργασίες μας. Ευχαριστούμε. Υπότιτλοι AUTHORWAVE